Λέω να αρχίσουμε τώρα. Δώσαμε ακόμα και ένα λεπτό παραπάνω. Σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω μία-δύο ανακοινώσεις από τη συνεδρία των συντονιστών, αλλά θα το κάνω προτού αρχίσει η ψηφοφορία. Τώρα προτείνω να εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης εξ ονόματος Επιτροπής της κυρίας Μακλάρκιν για το, την Επιτροπή Περιβάλλοντος που αφορά την ανακοίνωση Επιτροπής Αλληλεγγύη και Υγεία μειώνοντας τις ανισότητες στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πολύ ευτυχής που θα καλέσω τώρα την εισηγήτριά μας, την κυρία Μακλάρκιν, να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της και το χρονοδιάγραμμα και οποιοδήποτε άλλα θέματα θέλει να συζητήσει μαζί μας. Κυρία Μακλάρκιν, Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ αυτό το κρύο χειμωνιάτικο πρωινό. Θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα που αφορούν την ογνωμοδότησή μου, την οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Προσπάθησα να συμπεριλάβω ε, ό,τι μπορούσα με 1500 χαρακτήρες κάτι που δεν ήταν εύκολο εφόσον είχα να καλύψω τόσες πολλές πτυχές. Θα εστιαστώ σε αυτά που μπορούμε να προσθέσουμε ως Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών. Θελήσαμε να περιλάβουμε πράγματα όπως την, το, ε, τον τόπο κατοικίας των ατόμων, το κοινωνικό πλαίσιο, ε, επαγγελματική δραστηριότητα κλπ εγώ θέλω να τονίσω την ανάγκη προσπελασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας των φαρμακευτικών ε, θεραπείων που αποτελεί βασική πτυχή των ανισοτήτων στην τομέα της υγείας και επίσης ε, το θέμα της ε, διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης με βάση τη σχετική οδηγία. Όπως είπα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πιστεύω ότι οι πιο ουσιαστικές και πρακτικές προσθήκες που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτό το φάκελο αφορά τα επαγγελματικά προσόντα που καλύπτουν θέματα όπως αναγνώριση, αυτόματη αναγνώριση, κατανομή ε, και αλληλοενημέρωση για αυτό το θέμα, αλλά είναι σημαντικό να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές αρχές για να εξασφαλίσουμε τα προσωπικά πληροφορίες ανταλλάσσονται. Μιλούσα στη Βουδαπέστη σε επαγγελματίες υγείας σε μια διασυνοριακή ομάδα. Είναι οι ρυθμιστές των θεμάτων υγείας από όλες τις χώρες και νομίζω ότι αυτά τα συμπεράσματα τους μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμο στοιχείο. Συζητείται η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης κάτι στο οποίο αποδίδουν μεγάλη σημασία και το οποίο θα ήθελαν, θα ήθελαν να δημιουργηθεί. Ε, είχαμε και πρόσφατα δημοσίευση της έκθεσης κυρίας Εστρέλα που καλύπτει πολλούς άλλους σημαντικούς τομείς στους οποίους δεν είχα τη δυνατότητα να συμπεριλάβω. Τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση των μηχανισμών που θα περιορίσουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει βεβαίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις, υγειονομικ... τις δομές υγειονομικής που διαθέτουν χωρίς να παρέμβουμε σε αρμοδιότητές τους. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο, θα αναφέρω απλώς τώρα το χρονοδιάγραμμα. Οι τροπολογίες, ε, λίγη ημερομηνία κατάθεση των τροπολογιών στις 7 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η εξέταση θα γίνει από την Επιτροπή στις 10 Ιανουαρίου το απόγευμα μετά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές και λόγω αυτού αυτών των στενών περιθωρίων θα πρέπει να συνεδριάσουν οι σκιώδεις ηγητές στο Στρασβούργο αν αυτό είναι δυνατό. Ελπίζω σε Επιτροπή ΙΜΚΟ να συμβάλλουμε ουσιαστικά σε αυτό το νομοθέτημα. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές για να ακούσω τις απόψεις και τις θέσεις τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια και σίγουρα μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία τα οποία θα εμπλουτίσουν ε, <clears throat> την ε, έκθεση και όταν έγινε το, το συνέδριο διαπίστωσαν πόσο δεσμευμένοι είμαστε έναντι αυτού του θέματος και πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την αποφασιστικότητά μας στην Επιτροπή. Θέλετε <clears throat> να μιλήσετε, να λάβετε το λόγο παρακαλώ απευθύνουμε στα μέλη μας. Το ΕΛΚΑ ακόμα δεν έχει έρθει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Μακάρτη για τη γνωμοδότησή της η οποία σαν εργασία ε, ήταν κάτι το αρκετά δύσκολο. Εγώ θα συμβάλλω όσο μπορώ, γιατί στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Υγεία και Περιβάλλοντος έχω ασχοληθεί με τα θέματα της υγειονομική περίθαλψη. και πιστεύω ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο δεν αναφέρατε στο σημείο 1, Αναφέρεστε στα κοινωνικο-οικονομικά αίτια αλλά υπάρχουν και θέματα ε, χώρου, χωροταξίας και άλλα που πρέπει επίσης να υπογραμμιστούν. Βεβαίως ε, βρισκόμαστε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και έχουμε αναφερθεί στην παράγραφο 6 στην οδηγία για τις ε, υπηρεσίες για τα, για τα επαγγελματικά προσόντα πρέπει να προσέξουμε αυτή την παραπομπή γιατί στα θέματα της υγείας δεν πρέπει να θεωρήσουμε την υγεία σαν ένα εμπορικό προϊόν, σαν ένα εμπόρευμα, σαν τα άλλα. Γι' αυτό έχω κάποιες αμφιβολίες. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και η εσωτερική αγορά οπωσδήποτε και αναφέρομαι, δεν θυμάμαι πια σε ποια παράγραφο πρέπει να αναφερθώ, νομίζω στην 5 μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες υγείας στην υγειονομική περίθαλψη. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να πούμε ότι βεβαίω διατηρούν τι αρμοδιότητέ του τα κράτη-μέλη. Αλλά όπω βελτιώσαμε το κείμενο τη Κομισιόν στην ε, οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αποτελεσματική και θετική συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και υγειονομικής περίθαλψης επιμερίζοντας τις έρευνες, συμμετέχοντας σε κοινά δίκτυα, επιμερίζοντας επίσης το υλικό, το ιατρικό που κοστίζει ακριβά για χώρες που έχουν κοινά σύνορα όπως είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χρήματα και έστω και αν δεν εξαρτάται από την Επιτροπή μας τόσο πολύ να πούμε ότι μπορούν να γίνουν αυτές οι οικονομίες μέσα από έξυπνη και αποτελεσματική συνεργασία, αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων εκστρατιών ενημέρωσης των πολιτών για να συνηθίσουν σε καλύτερη προσωπική φροντίδα και υγεία. Διότι μόνο έτσι θα προστατεύσουμε και θα διατηρήσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας μας και πρέπει να παροτρύνουμε τα κράτη να οργανώνουν εκστρατείες πρόληψης όπως γίνεται σε ορισμένες χώρες και να προβλέπονται υποχρεωτικές εξετάσεις προληπτικές για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Και βεβαίως πρέπει να φροντίσουμε ιδιαίτερα και τα ηλικιωμένα άτομα διότι ο πληθυσμός της υπήρου μας γυρνάει και μήπως θα πρέπει να δημιουργήσουμε ειδικέ υπηρεσίες υγειονομικής περίθελψης, κατοίκων για τα ηλικιωμένα άτομα, ιατρικής περίθελψης αλλά και κοινωνικής φροντίδας υπηρεσίες αυτές που εξαρτώνται από την ε, Επιτροπή μας, ε, διότι αυτό είναι κάτι επίσης που θα δημιουργήσει ε, θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και θα δημιουργήσει χρήματα για τη διαφύλαξη του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ενώ καθημερινά θα βελτιώνεται η υγεία των ανθρώπων μέσα από υπηρεσίες που θα βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικία τους για τα επαγγελματικά προσόντα νομίζω ότι μπορούμε να σημειώσουμε ουσιαστικέ προόδου σε συνεργασία με τον Επίτροπο Μπαρνιέ, ο οποίος ε, ακολουθεί την ίδια γραμμή όπω εμά όπως και εμείς ε, με την επαγγελματική κάρτα και όλα αυτά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες, ειδικότερα για τα άτομα που δεν είναι πλέον σε θέση να τύχουν υγειονομική περίθαλψη, διότι δεν εντάσσονται πλέον στα συστήματα υγείας. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ανάλογο με αυτό που προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε ε, ε, ένα σύστημα οικουμενικής, οικουμενικής κάλυψης για τους ανθρώπους σε μέρες σαν και αυτοί που βρίσκονται στο δρόμο και χρειάζονται σε ιατρία, δωρεάν υπηρεσίες και σε κέντρα υγείας δωρεάν υπηρεσίες. Αυτό είναι οπωσδήποτε κάτι που υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υποχρέωση να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν τέτοιες υπηρεσίες που θα συμβάλλουν και στην αύξηση της απασχόληση. So, Ευχαριστώ. Μπερναντέτ, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Έχω Έχω μία ερώτηση να κάνω, διότι νομίζω ότι πρόκειται για ένα σφάλμα μεταφραστικό. 7 Δεκεμβρίου συζήτηση και 10 η ψηφοφορία, νομίζω ότι μάλλον είναι λάθος τυπογραφικό. 7 ε, Ιανουαρίου μάλλον θα εννοεί. 7, 7 Δεκεμβρίου για τα μέλη προθεσμία και 10 Ιανουαρίου είναι η πρώτη μέρα που θα επιστρέψουμε μετά τη διακοπή η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρούτσμαν. Εκ μέρου των συναδέλφων, ο κύριος Μπορζόινα, εκ μέρου των συναδέλφων, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακλάρκιν για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τους, κατανα... για τους πολίτες μας. Μιλάμε για την υγεία και ανισότητες που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Βέβαια, είναι ένα θέμα κοινωνικό ε, και διασυνοριακό, διότι αφορά ε, και την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών μας πέραν των συνόρων <clears throat> των εθνικών. Ε, αυτές οι ανισότητες λοιπόν θα πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες. Αυτό ορίζεται από τις συνθήκες υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι αναγκάζονται επειδή δεν υπάρχουν οι αντίστοιχε υπηρεσίες να μεταβούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και η Κομισιόν, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κομισιόν προωθεί αυτόν τον τομέα της ε, δρέωσης πλέον της ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη. Ε, έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις στον τομέα της υγείας τα επόμενα χρόνια, οι οποίες ε, θα οξύνουν ακόμα περισσότερο τις ανισότητες. Καταρχάς, πρόκειται για τις επιπτώσεις βεβαίως εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης και υπάρχουν πολίτες που αναγκάζονται να περάσουν μέσα από χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες και δεύτερον υπάρχει και το ο δημογραφικός παράγοντας ε, που πιέζει. Είναι λοιπόν ένα λίγο σημαντικό θέμα που, στο οποίο θα πρέπει να βρούμε ε, λύσεις. Η κυρία Μακλάρκιν απαντά ε, σε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα και θα ήθελα να συμπληρώσει τη γνωμοδότησή της με, μερικές, με μερικά ακόμα σημεία. Οι ανισότητες δείχνουν ότι χρειαζόμαστε μία διασυνοριακή απάντηση σε προβλήματα ε, τα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση. Η, ανισότητες ε, πρέπει να καταπολεμηθούν εκεί όπου δημιουργούνται, στην πηγή δηλαδή. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα του προσωπικού υγείας. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν έλλειψη στη χώρα μου, στη Ρουμανία, κυρία Μποντάνοβα οπωσδήποτε έχει υπόψη και την δική της χώρα, τη Βουλγαρία. Έχουμε προβλήματα προσωπικού και πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της κινητικότητας και να το ενισχύσουμε. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να ρυθμιστεί. Επίσης, ειδικέ περιπτώσεις, ειδική περίθαλψη από ιατρικές ειδικότητε. Εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα ωφελεί τους ασθενείς που χρειάζονται ειδική περίθαλψη με λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό δεν σημαίνει, εάν εφαρμόσουμε την επικουρικότητα, ότι δεν μπορούμε να λάβουμε καμία πρωτοβουλία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την συγγήτρια λοιπόν για τη γνωμοδότησή της. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Τσαλεμόσα, ο κύριος Κρούτσμαν, Κρούτσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Μακλάρκιν για την γνωμοδότησή της. Έχω ορισμένες, να προτείνω ορισμένες προσθήκες. Βέβαια το περιθώριο που έχουμε προτάσεων είναι λίγο περιορισμένο. Στο σημείο 4 αυτά τα οποία αναφέρει είναι πάρα πολύ καλά, είναι εξαιρετικά. Διότι εδώ μπορούμε να δράσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή συλλογή στοιχείων, ανταλλαγή στοιχείων, πληροφοριών ε, για την εξομάλυνση αυτών των ανισοτήτων. Επίσης το σημείο 8 είναι σωστό δεδομένου ότι και η Επιτροπή μας, η ΙΜΚΟ, έχει να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο όσο ασφαλά, όσον αφορά την ασφάλεια στον τομέα της υγείας και στα προϊόντα της. Ε, έχω ορισμένες επιφυλάξεις για το σημείο 3 όπου μιλάτε για την προσπελασιμότητα ε, και την προσιτότητα φαρμακευτικών θεραπείων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε ε, ποιο στοιχείο από τα δύο είναι πιο σημαντικό. Η πρόσβαση, η προσπελασιμότητα πιστεύω. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα, εκεί είναι η βασική πρόκληση εφόσον εξασφαλίσουμε ή βελτιώσουμε το θέμα της πρόσβασης, της προσπελασιμότητας, μετά μπορούμε να κοιτάξουμε την ε, προσιτότητα, το κατά πόσον δηλαδή οι θεραπείες αυτές είναι προσιτές. Η δυνατότητα πρόσβασης σε θεραπείες, η πρόσβαση, αυτό είναι το καθοριστικό σημείο. Εκεί αυτό πρέπει να τονίσουμε και ενδεχομένως να προσθέσουμε και κάτι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες της εσωτερικής αγοράς για πρόορες διαγνώσεις. για, προληπτικές, για προληπτική διάγνωση, συγγνώμη. Ε, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τα προβλήματα. Ε, σε αυτούς τους, στα δύο σημεία θα υποβάλω τροπολογίες. Κατά τα άλλα ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την θαυμάσια γνωμοδότηση. Ο κύριος Κρότσμαν τώρα, λέει ο πρόεδρος, έχει σειρά που περιμένει υπομονετικά. Ε, θα ήθελα και εγώ όμως προηγουμένως να προσθέσω μερικά σημεία. Και εγώ νομίζω ότι η κυρία Μακλάρκιν έχει ε, παρουσιάσει ε, μια θαυμάσια γνωμοδότηση η οποία σίγουρα θα περιέχει στοιχεία που προσθέτουν αξία στις εργασίες μας. Ε, όσον αφορά το έγγραφο της Κομισιόν, μου έκανε εντύπωση που δεν περιέλαβε το προσωπικό, το, το, προσωπικό υγείας, δεδομένου ότι η περαιτέρω εξέλιξη του, του προσωπικού υγείας ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να επιβάλλουμε μία ε, ισότητα υγειονομικής περίθαλψης. Πάρα πολλά προβλήματα προσπελασιμότητας ε, εξαρτώνται από την προσφορά εργασίας από τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερους επαγγελματίες υγείας. Άρα το θέμα αυτό δεν πρέπει να παραλυφθεί. Και θα υποβάλω τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση και κάτι άλλο που έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Πώς οι υπηρεσίες υγείας επενδύουν και πώς μπορούν να ενισχύσουν νέες καινοτομικές λύσεις, να προωθήσουν νέες καινοτομικές λύσεις, επενδύσεις και καινοτομίες. Ένας ε, επιτυχής συνδυασμός, αυτό χρειάζεται για την παροχή σωστών ε, υγειονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, ε, αλλά και σε ηλικιωμένους ανθρώπους, άτομα της τρίτης ηλικίας, στο να μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους, να έχουν τα κατάλληλα μέσα για να μπορούν να καλέσουν βοήθεια, για να μπορούν να αυτοβοηθηθούν. Δεν είχα κατανοήσει μέχρι τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόβλημα και η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει αργήσει πάρα πολύ να εκδώσει μια γνωμοδότηση σε αυτό το θέμα και, και εμείς ένα χρόνο για να προετοιμάσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Έχουμε τώρα βεβαίως μια έκθεση καινοτομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παρέχει πολλά νέα στοιχεία για να προωθηθούν οι καινοτομίες και επίσης συμφωνώ με την κυρία Σάλτε και ξέρουμε ότι θα υποβληθούν και περισσότερες γνωμοδοτήσεις για τη βελτίωση της φαρμακευτικής αγοράς και την ενθάρρυνση περαιτέρω επενδύσεων ε, για καινούργια φάρμακα και καινούργιες θεραπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά μου φαίνονται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και προς αυτό με αυτό το περιεχόμενο θα υποβάλω μερικές τροπολογίες. Εάν δεν θέλει κάποιος άλλος να παρέμβει. Α, ο κύριος Σεν από την Κομισιόν και μετά θα δώσω πάλι το λόγο στην εισηγήτρια να ολοκληρώσει. Ο κύριος Σεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να εκφέρουμε γνώμη επί του εγγράφου Καταρχήν, ένα, μια πρώτη παρατήρηση. Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης και της εφαρμογής της, ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία τα οποία τονίσαμε, για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε ό,τι φορά την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, είναι αυτό που ονομάσαμε health policies. Είναι γεγονός ότι προσπάθειες τόσο της Κομισιόν όσο και της δικής κοινωνικής επιτροπής είναι πολύ σημαντικές διότι η η υλοποίηση όλων των ε, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητε για να ασχοληθούμε με τα ζητήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πτυχή η οποία αφορά πολλές πτυχές. Πολλά, ε, πολλές πτυχές όπως κοινωνική, γεωγραφική, οικονομική κλπ. Επί των επιμέρους σημείων που αναφέρθηκαν να πω τα εξής. Αφενός ε, αυτό που τόνισαν οι διάφοροι αγορητές το ζήτημα της ε, κοινωνικής θέσης, κάτι το οποίο τονίζει και η Κομισιόν αλλά και πολλές μελέτες που έχουν κυκλοφορήσει, όπως η έκθεση Λαμορμότου για τον Βασίλειο, ε, υπάρχει και μια γεωγραφική πλευρά του προβλήματος, διότι η ανισότητα στον τομέα της υγείας είναι κάτι το οποίο τονίζεται συχνά ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να ξεχνάμε και τις ανισότητες που υπάρχουν και στο πλαίσιο του ιδίου κράτους και ανάμεσα σε περιφέρειες ε, και έχω κατά νου κράτη τα οποία έχουν εκτεταμένη εδαφική κάλυψη Α, υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορές ανάμεσα σε περιφέρειες ε, στο ίδιο κράτος μέλος, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις αστικές περιοχές και στις ε, αγροτικές περιοχές. Την Ήπεθρο. Τώρα, σε ό,τι φορά την υλοποίηση αυτής της ανακοίνωσης, η ανταλλαγή στοιχείων και εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό η η Κομισιόν το τονίσει περαιτέρω σήμερα, ότι δηλαδή η ανταλλαγή δεδομένων είναι θεμελιώδες θέμα. Βελτιώνουμε τις γνώσεις μας ε, μέσω της ε, ανταλλαγής ε, δεδομένων στα θέματα υγείας και σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Οι υπηρεσίε Κομισιόν εργάστηκαν εντατικά του τελευταίου μήνε, αφενό για να βελτιώσουμε τι γνώσει μα και αφετέρου για να υλοποιήσουμε και αυτό θα συμβεί μέσα στους προσεχείους μήνες, όπως εξάλλου είχε προβλεφθεί και στο κείμενο της ανακοίνωσης, να εφαρμόσουμε μια σειρά δικτών που προτείνονται στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας προκειμένου να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των θεμάτων της ανισότητας στον τομέα της υγείας. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Oh, sorry. Ευκαιρία ε, ανταλλαγή απόψεων στην ε, Επιτροπή μας για το ζήτημα των δικτών και των διαφορών ανάμεσα στις Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μακλάρκιν προκειμένου να ολοκληρώσει ε, και αν έχει να κάνει κάποια σχόλια. Κυρία Μακλάρκιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να θίξω μερικά σημεία. Ο Μπολτζόη από το Άλντε ε, τόνισε πόσο σημαντικό είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες και για μας ως πολίτες και νομοθέτες να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανισότητε που υπάρχουν στο τομέα τη υγεία και αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι μια προτεραιότητα για τους πολίτες μας, άρα αποτελεί προτεραιότητα και για μας. συμφωνα απόλυτα με το ότι η ιστορική αγορά, η Επιτροπή Ιστορική Αγοράς θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτήν την ανακοίνωση, διότι η αγορά δεν ε, μπορεί να βοηθήσει, αλλά και εμείς ε, από πλευρά μα μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, να δημιουργήσουμε αυτό το κινητό περιβάλλον που απαιτείται, προκειμένου να εξευρεθούν καλύτεροι τρόποι περίθαλψη και θεραπεία μέσω των αγορών. Τώρα, για κυρία Σόλντε Μόζερ, ναι, πιστεύω ότι η θεμελιώδη ε, περίθαλψη είναι ένα πολύ σημαντικό, θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ανταλλαγέ ε, βέλη των πρακτικών Φυσικά χρειάζεται να λαμβάνουμε όλε τι απαραίτητε πληροφορίε και να τι ανταλλάσσουμε. Εντάξει, τα σημείωσα όλα τα σχόλιά σα και θα τα λάβω υπόψη μου. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλε, βλέπω πω ε, έφτασε. Ξέρω ότι συνεργάζεται με την κυρία Μακλάρκιν. Απλά ήθελα να σημειώσω πως ε, φράσατε ανάμεσά μας. Έχετε το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Μακλάρκιν θα εξετάσει τροπολογίες σας. Δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία να συζητήσουμε το ζήτημα πριν από τον Ιανουάριο. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια σύντομη ε, συζήτηση επί των τροπολογιών. Η κυρία Μακλάρκιν θα συναντήσει τους γεώδεις συγητές ενδεχόμενα στο Στρασβούργο για να συνεργαστούν. Ευχαριστώ την Κομισιόν και τώρα... Επόμενο σημείο είναι οι ψηφοφορίε στις 10 η ώρα. Ας διακόψουμε λοιπόν για μερικά λεπτά προκειμένου να μπορέσουν να προετοιμαστούν οι πολιτικές ομάδες και στις 10 ακριβώς ε, ξεκινάμε τις ψηφοφορίες.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

Uh, Ωραία λοιπόν κυρίες και κύριοι Είμαστε έτοιμοι για τις δύο ψηφοφορίες που έχουμε σήμερα το πρωί Καλημέρα σε όλους Χαίρομαι που έχουμε μια καλή παρουσία μελών εδώ παρόλο τον καιρό. Είχαμε μια πολύ καλή συνεδρίαση και μια πολύ καλή συζήτηση με την έκθεση της κυρίας Μακλάρκιν και η γνωμοδότηση αυτή θα ψηφιστεί στις 10 Ιανουαρίου. Δυστυχώς δεν ήταν κανείς κοιόδης από το ΕΛ, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλουν με τροπολογίες στη συζήτηση. Τώρα που είμαστε όλοι εδώ θα ήθελα να σας ενημερώ, ενημερώσω για τις αποφάσεις που πήραμε χτες τους συντονιστές διότι δώσαμε μερικές θα αναθέσαμε μερικές εκθέσεις και τις θα τις περάσω γρήγορα. Λοιπόν, ε, θα αναλάβουμε ορισμένες μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις Καταρχάς, για, στο 2-3 ευρωζωνική θα γίνει από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς το Ευρωπαϊκό Συμβατικό Δίκαιο θα πάει στο ΕΛΚ. Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Επαγγελματική Κατάρτιση στους σοσιαλιστές, οι καινοτομίες θα γίνει από την GUE NGO και το 2.7 ε, προϋπολογισμός θα, γίνει από το ΕΛΚ και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανδώρα θα γίνει από την ομάδα ΑΛΤΕ το 2.8. Ωραία, ε, θα αναθέσουμε λοιπόν την εργασία στους εισηγητές σύντομα και θα ξεκινήσει η δουλειά και επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών έχει ε, παραταθεί μέχρι τις 26 Ιανουαρίου. Η κυρία Στάιλερ θα αρχίσει τις ε, διαβουλεύσεις σήμερα, αν είναι εδώ οι συντονιστές της έδωσαν εντολή να διαβουλευθεί για τη δεύτερη ανάγνωση με το Συμβούλιο στα θέματα τα κατασκευαστικά, κατασκευαστικά έργα για το φόρουμ της ενιαίας αγοράς που θα είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, πιο φιλόδοξο από το πιλωτικό η κυρία Τούν, Χέρνσταν και Μπουζόη και οι κυρίες ε, θα συμμετάσχουν στην Οργανωτική Επιτροπή και θα συναντηθούμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά θέματα, αλλά βεβαίω θα σταλεί και μία, ένα επίσημο σημείο σε όλα τα μέλη αφού εγκριθεί από τους συντονιστές. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ο κύριος, η κυρία Βάσμπεργκερ είναι εδώ και μας ζήτησε αν μπορούμε να ψηφίσουμε καταρχάς την έκθεση της κυρίας Βάιλερ και όσον αφορά το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου έχετε ένα αντίγραφο της τελικής θέσης το οποίο μας, την οποία μας έστειλε το Συμβούλιο με επιστολή που λέει ότι είναι πρόθυμοι να τη δεχτούν. Επίσης μια ανακοίνωση Κοινοβουλίου Κομισιών ε, που συνοδεύει αυτήν την, τον τριμερή διάλογο. Θα δώσω λοιπόν ε, καταρχάς το λόγο στην κυρία Βάις Γκέμπερ για να ζητήσω την έγκρισή σας. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχάς θέλω να πω ότι με αυτήν την έκθεση την οποία ελπίζω να έχουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον έχουμε προχωρήσει ένα βήμα. Θέλουμε τώρα να μεταφράσουμε τις προτάσεις σε έργα και να ε, ολοκληρώσουμε το θέμα των πινάκων, των ε, correlation tables. Αυτοί οι πίνακε σχέση ακόμα κρεμούν, αλλά έχουμε βασική συμφωνία από αυτών. Και ευχαριστούμε το Συμβούλιο που μας βοήθησε στις εργασίες μας και ευχαριστώ και τον πρόεδρο της διάσκεψη των, ε, ευχαριστώ τον πρόεδρο ο οποίος στη διάσκεψη των πρόεδρων συνεχώς μας ε, ε, ενίσχυσε στη θέση μας και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει απλώς για αυτήν την έκθεση η οποία είναι πάρα πολύ τεχνική όπως το είπε και η κυρία Ρούλε την περσμένη εβδομάδα δεν μπορέσαμε να βρούμε μια εντελώ διαφορετική διατύπωση. Εν πάση περιπτώσει μπορέσαμε να βρούμε μια διατύπωση αυτών των πινάκων ε, αντιστοιχειών που, ε, επί των οποίων πιστεύω θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Αυτοί λοιπόν οι πίνακες πιστεύω να εγκριθούν διότι τις έχουμε μελετήσει ιδιαίτερα και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι με αυτήν την γραμμοδότηση θα μπορέσουμε να μειώσουμε το βάρος της γραφειοκρατίας Ταυτόχρονα δε να επιτύχουμε μια οριζόντια, έναν οριζόντιο συντονισμό αυτών των ε, πινάκων αντιστοιχίας, ε, των correlation tables. Όπως σας είπα, το ντοσιέ αυτό είναι πάρα πολύ τεχνικό και δεν υπάρχουν διαφορές απόψεων πλέον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βάις Γέρμπερ. Όπως είπατε το θέμα αυτό είναι περίπλοκο, αυτοί οι πίνακες αντιστοιχειών έχουν συζητηθεί επί μακρόν, τελικά από το Μάιο πιστεύω ότι τώρα φτάσαμε στην τελική φάση και να... ότι θα προχωρήσουμε ικανοποιητικά. Δεν ξέρω εάν επιθυμεί να μιλήσει και ο εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είμαστε ικανοποιημένοι με, την τελική, με το τελικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είχαμε πολύ επικοδομητικές διαβουλεύσεις. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη συνεργασία της. Πραγματικά είχαμε καρποφόρες και επιτυχείς ε, συζητήσεις που κατέληξαν σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σε αφορά την ανακοίνωση, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν, διότι ο κύριος Στάινερ ήταν εδώ πριν από δύο εβδομάδες και μίλησε ότι θα υπάρχει του χρόνου μια νέα πρόταση για, την, για τα όργανα μετρολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν τι έχει να μας πει επ' αυτού. Η Κομισιόν στην ανακοίνωση, όπως λέει, ε, θα κάνουμε αυτήν την αναθεώρηση. Θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια διαδικασία για αυτά τα θέματα όπως και στο παρελθόν. Right. Πολύ ωραία. Υπάρχει λοιπόν μία πρόταση να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα όσοι λοιπόν είναι υπέρ αυτής της θέσης πρέπει να μετρήσουμε. διότι πρέπει να καταχωριστούν ε, οι ψήφοι και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες. Κατά. Αποχές. Πολύ ωραία ομόφωνα με 32 ψήφους εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε πολύ. So um, Βάις Γκέρμπερ. Θα φροντίσουμε λοιπόν uh, make... θα φροντίσουμε ότι θα καταχωρηθεί για ολοκληρωμένη συζήτηση στην Ολομέλεια δεν ξέρω αν κάποιος φροντίστε να ζητήσετε ε, επαρκή χρόνο ε, κυρία Βάις Γκέρμπερ, για να έχουμε τη δυνατότητα για μια συζήτηση. Θα ψηφίσουμε τώρα για το δεύτερο θέμα, που είναι η γνωμοδότηση της κυρία Βάιλερ για τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων. Έχει γίνει όλη η δουλειά με τους Σκιώδης, ήμουν εκεί χθες Μπάρμπαρα Βάιλερ, θα μας πείτε δύο-τρία πράγματα πρωτού ψηφίσουμε. das kann ich Πολύ σύντομα. Συζήτησα χτες με τους συζητητές. Έχουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 1, την οποία διατυπώσαμε μαζί. η οποία πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό και λογικό το περιεχόμενό της και εκτός από τους πράσινους έχω την, επιβεβαίωση ότι οι άλλοι θα δεχθούν την συμβιβαστική τροπολογία Ένα, Πιστεύω ότι οι πράσινοι δεν είχαν λόγω, είχαν λόγω καιρού προβλήματα και δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν μαζί μου. <clears throat> Πιστεύω ότι έχουμε μία γνωμοδότηση στην οποία θα μπορέσουμε να την υπερψηφίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία. Λαμβάνουμε υπόψη, έχουμε λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων και όλων όσοι, όσων ασχολήθηκαν με το θέμα της, ε, ε, των επιπτώσεων, της, της μελέτης επιπτώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Δεν... Επειδή είναι σύντομη η ψηφοφορία, θα ψηφίσουμε με ανάταση της χειρός. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες. Παράγραφος 2α. Κρόιτσμαν. Υπέρ. Να μετρήσουμε, θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθως. 20, 20. So that's, uh, so that's going to pass anyway, 20 in favor. Um, those against. Κατά. That's carried then. Δεκτό. 20 έναντι 12. Τροπολογία 3 με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, δεκτή. Καταπίπτει η 3, 4 Κρόιτσμαν υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 5 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 6 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Δεκτή. Καταπίπτει 6 Κρόιτσμαν, συμβιβαστική τροπολογία υπέρ, κατά, δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 9, Κρόιτσμαν, υπέρ, κατά, δεκτή, σαφώς δεκτή. 10 Κρόιτσμαν, υπέρ, κατά, δεκτή. Τροπολογία 11 Κρόιτσμαν υπέρ, κατά, απορρίφθηκε σαφώς. 13 Κρόιτσμαν υπέρ, κατά, δεκτή. 14 υπέρ, κατά, δεκτή. Και σε ό,τι αφορά τη 15, νομίζω ότι κάτι θέλει να πει η κυρία Βάιλερ. Θα πρότεινα μια μικρή προφορική τροπολογία για να ικανοποιήσω την εισηγήτρια. Έχουμε διπλοποίηση, επανάληψη στη διατύπωση. Καταργώ λοιπόν τις λέξεις και των κρατών μελών στο 9, να το διαβάσω. Τονίζει ότι οι ρυθμίσεις Έξυπνη νομοθεσία με βάση την πλήρη και αντικειμενική εκτίμηση επιπτώσεων παραμένει κοινή ευθύνη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και Οργάνων και ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεκτιμά τι αντιδράσει που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Νομίζω αυτό ικανοποιεί την εισηγήτρια. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Citations Κρότσμαν, οπότε θα ψηφίσουμε τώρα για το σχέδιο γνωμοδότηση στο σύνολό του. Υπέρ. Είναι κάποιο κατά. Ομόφωνα. Δεν είχαμε και αποχέ, ομόφωνα δεκτή λοιπόν. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια κυρία Βεβαίω θα χρειαστεί να γίνει περαιτέρω δουλειά η κυρία Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε γιατί θα περάσει, θα πάει στην Ολομέλεια νομίζω μόνο το Μάρτιο. Όχι νωρίτερα. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για όσους δεν θα παραμείνουν στην αίθουσα και προτού περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η οδηγία, μάλλον ο κανονισμός για την έγκριση αγροτικών και δασικών οχημάτων. Ο κύριος Παντσέρη είναι εδώ και σύμφωνα με τις αρχές που, συνεφώνησαν, που συμφωνήθηκαν μεταξύ των συντονιστών, σύμφωνα με αυτά που συμφωνήσαμε στη συνεδρίαση των συντονιστών, θα ξεκινήσει η συζήτηση με μία παρουσίαση της ε, ε, αξιολόγησης επιπτώσεων από την Επιτροπή θα παραδώσω τη θέση μου στον Αντιπρόεδρο Νιού γιατί θέλω να συμμετάσχω, θέλω να συμμετάσχω ως σχεώδης εισηγητής της συζήτηση στις, ε, στις 11 και 4 θα πάω στην Επιτροπή των Περιφερειών για... και γι' αυτό θα δώσω το λόγο αμέσως στην Αντιπρόεδρο η οποία θα αναλάβει από εδώ και πέρα την Προεδρία της συνεδρίασής μας.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 Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Όλοι έχετε παραλάβει το έγγραφο που διανεμήθηκε και επειδή είμαστε ακόμα μέσα στα χρονικά περιθώρια, επειδή θέλουμε να υπάρξει και καιρό για συζήτηση, θα δώσω αμέσω το λόγο στην Επιτροπή, η οποία θα μα παρουσιάσει το έγγραφο που μόλι σα διανεμήθηκε για τι επιπτώσει και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάκομο Ματίνο. Σα αφήνω χρόνο να καθίσετε, να οργανωθείτε. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους γιατί δώσετε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την αξιολόγηση επιπτώσεων των νομοθετικής πρότασης για τα, τους ελκυστήρες, τους δασικούς και τους αγροτικούς. Πρόκειται για νομοθεσία πλαίσιο και προτού αφιερώσω λίγο χρόνο στην παρουσίαση, θα ήθελα να σας θυμίσω το ευρύτερο πλαίσιο αυτής ε, της πρότασης. Όπως ξέρετε, ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προβεί σε μια ε, επικαιροποίηση και απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι που έχει γίνει για τα ιδιωτικά, για τα επιβατικά αυτοκίνητα από το 2007 και μετά το 2009 με τη Γενική Νομοθεσία για την Ασφάλεια. Και τώρα έχουμε διατυπώσει μία πρόταση που θα καλύψει άλλες άλλους δύο πολύ σημαντικούς τομείς, τα, τα, τους αγροτικούς και δασικούς ελκυστήρες που θα συζητήσουμε σήμερα το πρωί, ενώ το απόγευμα με τα μεγάλη χαράς θα βρίσκομαι και πάλι εδώ, διότι θα γίνει μια παρουσίαση της αξιολόγησης επιπτώσεων για τις ε, μοτοσυκλέτες και τα άλλα συναφή οχήματα. Στη διάρκεια της εξέτασης ε, θα δούμε ότι θα χρειαστεί να αλλάξουν, να είναι διαφορετικές ορισμένες διατάξεις. Αλλά τα δύο μέτρα είναι σημαντικό να ενταχθούν στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο με σκοπό την απλούστευση της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου. Θα σας δείξω τώρα με τη βοήθεια μερικών διαφανειών το συλλογισμό πάνω στον οποίο βασίστηκε η αξιολόγηση επιπτώσεων. Στη νομοθεσία αυτό που καλύπτουμε είναι η έγκριση τύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξίζει να θυμίσουμε ήδη από τώρα ότι δεν είναι κάτι το καινούριο, είναι κάτι που συνυπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις με τις εθνικές εγκρίσεις τύπου, αλλά υπάρχει μια προστιθέμενη αξία, διότι οι κατασκευαστές των οποίων τα προϊόντα φέρουν τον τύπο, ε, τον, ε, την έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να, να διοχετεύουν τα προϊόντα τους σε, στο σύνολο της αγοράς. Αυτό δεν είναι κάτι το νέο, υπήρχε και στο παρελθόν. Αλλά στην περίπτωση των αγροτικών και δασικών ελκυστήρων, ένα κρίσιμο στοιχείο ήταν η κάλυψη της ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου για τις διάφορες κατηγορίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που χρειάζεται να καλύψουμε με μεγάλες διαφορέ. με σημαντικές διαφορές. Έχουμε τους ελκυστήρες που χρησιμοποιούν ε, έχουμε πολύ μικρούς, περνάμε από τους πολύ μικρούς ελκυστήρες σε μεγάλους, ε, πολύ ισχυρούς ε, μεγάλ, ε, με μεγάλης ισχύος Γι' αυτό το λόγο υπήρχε ανάγκη να εξορθολογήσουμε αυτόν τον τομέα και, τα διάφορα, και, τις, διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της, έγκρισης, της ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου δεν είναι ιδανική λύση για όλες τις κατηγορίες. Θα υπάρξει λοιπόν μια διαμόρφωση ώστε να έχουμε ε, πιο συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων για να ανταποκριθούμε στις ε, απαιτήσει και στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μια τοπική ή περιφερειακή παραγωγή και για τις οποίες ε, ε, η, έγκριση, η ευρωπαϊκή έγκριση τύπου να μην είναι πάντοτε απαραίτητη. Γι' αυτό θα διατηρηθεί και η εθνική έγκριση τύπου και θα υπάρχει στον, για τον κατασκευαστή η δυνατότητα επιλογής. Μιλάμε λοιπόν για κάτι το προαιρετικό. Επόμενη διαφάνεια όπως σας είπα σε ορισμένες περιπτώσεις η έγκριση τύπου θα είναι προαιρετική και παρόλο που υπάρχει ατομική έγκριση, μεμονωμένη έγκριση ε, τύπου οχημάτων δεν συνιστούμε ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή έγκριση τύπου για, αυτά, για αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Όπως ε, σας είπα και προηγουμένως, αυτό που θέλουμε να καλύψουμε είναι ε, μια απλουστευμένη ε, διαδικασία. Έχουμε την οδηγία πλαίσιο του 2003 συν 24, 24 ε, συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμογής οι οποίες έχουν δεχθεί πολλές ε, τροποποίησεις ε, ε, ώστε να ανταποκρίνονται και να παρακολουθούν τις τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Βεβαίως, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών καλούνται να ενσωματώσουν αυτές τις οδηγίες, να τις ενσωματώσουν σωστά στην εθνική τους νομοθεσία. Και ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκα είναι ήδη προηγουμένως είναι ότι το παρόν, το σημερινό πλαίσιο είναι πολύ περιορισμένο από πλευράς κάλυψης των εγκρίσεων τύπου. Και γι' αυτό θέλουμε να δούμε και εξετάσουμε πολύ προσεκτικά πώς θα επεκτείνουμε αυτή την έγκριση τύπου σε άλλα προϊόντα ειδικό, πέραν των δασικών και αγροτικών ελκυστήρων στα τρέιλερ, ε, στα ρημουλκά και τα ρημουλκούμενα. Μια ιδέα η οποία δεν εμφανίζεται στο κείμενο που έχετε μπροστά σας είναι η επικαιροποίηση των κανόνων ασφαλείας, ειδικότερα εκείνων που αφορούν τα φρένα, την πέδηση και άλλα στοιχεία που, έχουν, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων έγινε πριν από αρκετό καιρό. Το σχέδιο πρότασης είχε υποβληθεί πριν από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων έγινε το 2008 και το 2009 μετά από τη δημόσια διαβούλευση που έγινε και αυτή το 2008. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων και στην αξιολόγηση επιπτώσεων ε, καλύψαμε τους βασικούς πυλώνες. Την απλούστευση, την καλύτερη νομοθεσία, το γεγονός ότι τώρα προτείνουμε και αυτό είναι κάτι πρόσφατο έναν κανονισμό έγκρισης τύπου αντί ε, οδηγίας με μέτρα εφαρμογής αυτό που ονομάζουμε split level approach για να δούμε τι κάλυψη θα έχουμε ε, για τις διαφοροποιημένες κατηγορίες τι είδους έγκριση τύπου πρέπει να προβλέψουμε και αν χρειάζεται και αν πρέπει αυτή η έγκριση τύπου η ευρωπαϊκή να είναι υποχρεωτική ή σε ορισμένες περιπτώσεις να αφήσουμε, να διατηρήσουμε τις εθνικές εγκρίσεις τύπου όπως ισχύουν αυτή τη στιγμή. Επόμενη διαφάνεια. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης σε ό,τι αφορά τις άλλες κατηγορίες, ε, τις μοτοσυκλέτες ε, ειδικότερα, σε αυτή τη φάση δεν έχουμε αποφασίσει να επιφέρουμε σημαντικές μεταβολές στις τεχνικές απαιτήσει και προϋποθέσεις παρόλο που σε ορισμένους τομείς όπως είναι το σύστημα πέδησης στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες επικαιροποίησεις αλλά αυτά θα καλυφθούν καλύτερα από τη γνωμοδότησή μας σε ό,τι αφορά τα μέτρα εφαρμογής σε περαιτέρω δηλαδή νομοθετικά κείμενα δεν θα αλλάξουμε ε, δεν θα αλλάξει το περιεχόμενο των τεχνικών απαιτήσεων, διότι η αξιολόγηση επιπτώσεων συμμετείχαν οι καταναλωτές, η βιομηχανία και οι, τα κράτη-μέλη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δηλαδή και ε, εκφράστηκαν όλοι και είπαν ότι δεν χρειάζεται επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτήσεων διότι οι ισχύουσες παραμένουν ικανοποιητικές. Θα σας δείξω τώρα γρήγορα τις επόμενες διαφάνειες για, να μην χάνουμε χρόνο. Λίγα λόγια για το, τη νομική, νομοθετική νομική δομή. Κρίναμε ότι ήταν σκόπιμο να επιλέξουμε έναν κανονισμό που θα αντικαταστήσει την παρούσα οδηγία πλαίσιο έναν βασικό κανονισμό που θα περιλαμβάνει τρία ή τέσσερα τμήματα που θα καλύψουν τα θέματα της ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και τις διοικητικές διατάξεις. Η αξιολόγηση επιπτώσεων μας έδειξε επίσης ότι στο μέτρο του δυνατού και αυτή είναι μια τάση που τη βλέπουμε σε όλη την νομοθεσία ευρωπαϊκής έγκρισης τύπου ότι είναι καλύτερο να αναφερόμαστε σε διεθνή τεχνικά πρότυπα κάθε φορά που αυτά είναι διαθέσιμα και αυτό είναι συμβατό με το θέμα της, της ύψης της ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που θέλουμε να ε, εξασφαλίσουμε Η αξιολόγηση επιπτώσεων στην αρχή μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος η, μόνη, ε, η υποχρεωτική ευρωπαϊκή έγκριση τύπου δεν είναι κάτι το αναγκαίο για όλες τις 45 κατηγορίες Οπωσδήποτε χρειάζεται ένας, όμως ένας εξορθολογισμός όλων των κατηγοριών. Όπως είπα και προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι το θέμα της split level approach. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που αναφερόμαστε σε αυτό ή που συνιστούμε την ε, εφαρμογή αυτής της συγκεκριμένης προσέγγισης το συμπέρασμα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι το να χρησιμοποιήσουμε έναν κανονισμό μαζί με ένα σύντομο αριθμό ε, μέτρων εφαρμογή είναι η πιο αποτελεσματική και η πιο λογική προσέγγιση και απόλυτα παράλληλα συμβατή με τις προσεγγίσεις που εφαρμόζουμε για τις εγκρίσεις τύπου Τώρα μπορούμε να δούμε εντάχει τις επόμενες διαφάνειες. Α, εδώ κατά εξουξοδότηση πράξης. Υπάρχει ο κανονισμός για τη συναπόφαση που αποτελεί και το αντικείμενο της πρότασης. Στις ε, πράξεις εφαρμογής η ιδέα, η σκέψη είναι να συμπεριλάβουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές απαιτήσεις, και τις εναρμονισμένες διοικητικές απαιτήσει, διαδικασίες δοκιμών έντυπα για την ευρωπαϊκή έγκριση τύπου που πρέπει να είναι εναρμονισμένα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τις κατευθυνότητες πράξεις και το άρθρο 90 από τις πράξεις εφαρμογής βάσει του άρθρου 291 και στην πρότασή μας έχουμε προβλέψει τις σχετικές διατάξεις που θα εξουδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, θεσπίζει αυτού του είδους των πράξεων όποτε απαιτείται. Επόμενη διαφάνεια, νομίζω ότι τελειώνουμε. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η νομοθεσία συναπόφασης η οποία σαφώς ορίζει και περιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τις κατεξουδότηση και τις πράξεις και τις πράξεις εφαρμογής. Αυτό είναι περιττό να σας το θυμίσω, να σας το πενθυμίσω, αλλά όταν ακολουθούμε αυτή τη split level approach είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε από την αρχή αυτά τα στοιχεία. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τώρα σε ό,τι φορά την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, όντως αποτελεί πρόκληση σε αυτόν τον τομέα όπως και σε άλλους ε, υποθέσεις, σε περιπτώσεις που αφορούν οχήματα. Το split level approach θα πρέπει να συμβάλλει στο να υπάρξει μια πιο έγκαιρη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. Όπως προανέφερα, έχουμε διεθνείς και προ, διεθνείς αποφάσεις ε, και ε, πρότυπα από τον ε, ΟΣΑ. Έχουμε και τα πρότυπα και ΣΕΝΕΛΕΚ. ΑΙΖΟ και την ΣΕΝΣΕΝΕΛΕΚ. και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα CARS 21 που αποτέλεσαν μια στρατηγική επιρροή της ε, νομοθεσίας που αφορούν τον τομέα των οχημάτων. Έχουμε λοιπόν αυτά τα διεθνή πρότυπα τα οποία είναι απόλυτα συνεπή με τις ε, επιλογές μας. τα σε ό,τι split level approach, μια σειρά, προλέγουν μια σειρά από πράξεις κατεξιοδότηση που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας περιβαλλοντικές απαιτήσεις αλλά και εφαρμοστικές πράξεις που αφορούν στις διοικητικές ε, απαιτήσεις Τώρα, για να συμπληρώσουμε το σύνολο της νομοθεσίας υπάρχει και κάποια άλλα νομοθετήματα που αφορούν την περίοδο μέχρι τον Ιανουάριο 2014. Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, εκτός αν το επιθυμείτε, αλλά για να εξοικονομήσουμε χρόνο, να σταματήσω στο σημείο αυτό την παρουσίασή μου και να μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες, αλλά στην πρόταση αυτή, όπως είπα, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με νέες απαιτήσει, αλλά περιέχει τις βασικές απαιτήσει οι οποίες ε, αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα, διάφορα στοιχεία. Θα ήθελα ε, την ευκαιρία αυτή να πω ότι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τομέα των σε αυτοκινητομηχανίας ε, ε, των ελκυστήρων ε, αντιμετωπίζει μάλλον αντιμετωπίζεται με έναν κατακαιρματισμένο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο συνιστούμε την ε, πρόταση η οποία σας ε, γίνεται μέσω αυτού του κανονισμού, διότι είμαστε πεπισμένοι ότι αυτός ο κανονισμός θα φέρει εξορθολογήκευση του τομέα και θα αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις με άλλα νομοθετήματα, όπως παραδείγματος χάρη ε, θυμίστε πως υπάρχει το θέμα της αλληλεπικάλυψης με τον νομοθεσία περί μηχανών και μηχανημάτων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να έχουμε ένα πιο εξορθολογισμένο κείμενο. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι ελκυστήρες μπορούν να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμόγης οδηγίας ε, περί μηχανημάτων και οι ενδιαφερόμενοι, οι εμπλεκόμενοι, οι εθνικές αρχές και οι εφαρμοστικές αρχές τα κράτη-μέλη και οι κατασκευαστές θα, ε, θα μπορούν να εποφελθούν αυτοί από αυτήν την ε, μονοευθυντική σειρίδα που τους προσφέρεται σε ό,τι φορά την κανονισμό αυτών και την εφαρμογή του. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μαρτίνο για την παρουσίασή σας. Φυσικά μπορεί να μην είναι απόλυτα αναλυτική, αλλά μας δίνει μια πλήρη εικόνα. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν είχαμε θίξει μέχρι τώρα, αλλά πιστεύω πως ο εισηγητής μας Αντώνιο Παντσέρη θα μας ε, πει την ε, γνώμη του. Έχει δουλέψει πολύ επί του θέματος. Ε, θα δώσω το λόγο στον αγαπητό Αντώνιο και προτείνω δεδομένου ότι ο κύριος Μάντερς ε, θα απουσιάσει να δώσω μετά το λόγο στο ΕΛΚ, μετά στους πράσινους, ε, μετά στην ΓΟΕ και λοιπά και αν επιστρέψει ο κύριος Μάντερς θα πάρει το λόγο στο τέλος. Αντώνιο, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για μια εργασία την οποία έχουμε ξεκινήσει ε, και πρόκειται να την εμβαθύνουμε περαιτέρω στο μέλλον. Αυτό το οποίο μπορώ να πω σε αυτή τη φάση είναι πως ε, χρειάζεται να συμφωνήσουμε με την πρόταση διότι όλες οι διαδικασίες που οδηγούν σε εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς στην περίπτωση αυτή την έγκριση αναφορικά με αυτόν τον τύπο οχημάτων είναι μια τάση γενική και το Κοινοβούλιο θα πρέπει αλλά και η Ευρώπη συνολό τους να εργαστούν για να επιτύχουν με αυτόν τον στόχο. Έχουμε λοιπόν μια πρόταση η οποία τίνει να ε, συμπληρώσει, να βελτιώσει και να εξυγχρονίσει το ισχύον πλαίσιο δίνοντας ε, και ένα νομοθετικό πλαίσιο πιο συνεπές ε, τώρα. μετά από όσα άκουσα νομίζω πως θα πρέπει να μας δώσει κάποιες διαφορετικές η Κομισιόν για να μπορέσουμε να έχουμε μια προσέγγιση το δυνατόν συνενετικότερη τώρα. Οι διευκρινήσεις που θέλω να αναφέρω είναι ότι η επιλογή ενός γενικού κανονισμού και όχι κλαρικών κανονισμών που συνδέονται με τα διεθνή πρότυπα ε, θέτει το ερώτημα το πώς ε, μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές και αυτές οι τροποποιήσεις ε, Ρωτάω λοιπόν αν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με τρόπο αυτόματο ή κάτω από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα σε ό,τι φορά τους κλαδικούς κανονισμούς και την διαδικασία των πράξεων κατευθυνσιοδότηση θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι ο ρόλος και πώς μπορεί να επέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και ιδέες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ποιο είναι το πεδίο δυνατοτήτων που ανοίγεται για το Κοινοβούλιο τόσο σε ό,τι φορά την ολοκλήρωση της τουρκικής αγοράς και την εφαρμογή της. Πιστεύω ότι χρειάζεται να προστατεύσουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά και στην υπερεθνική αγορά δίχως να υπάρχουν διακρίσεις και ε, παροτρύνοντας την ε, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προκειμένου να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας διότι το ζήτημα της έγκρισης δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις ε, επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει και στο περιβάλλον και στην ασφάλεια αλλά και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ε, απασχόλησης και νομίζω ότι δεν λέγονται επαρκή πράγματα σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής για όλη την κατηγορία των οχημάτων σχετικά με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των ε, εργαζομένων. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα επί του οποίου χρειάζεται να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω. Τέλος, να ρωτήσω αν υπάρχουν ε, διστάμενες απόψεις ε, από τους ενδιαφερόμενους ε, αν υπάρχει μια συζήτηση γραμμικού χαρακτήρα ή αν έχουν τεθεί και άλλες εναλλακτικές λύσεις και κάτι ακόμα. Η εκτίμηση αντικτύπου δεν εξηγεί όλες τις αλλαγές που έγιναν στο νομοθετικό, στο κανονιστικό πλαίσιο και ως εκ τούτου πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκινήσει λίγο παραπάνω όλα αυτά τα στοιχεία αλλά και τα θέμα των κατευθύντων πράξεων αλλά και των εφαρμοστικών πράξεων και αν υπάρχει κάποιες προθεσμίες, κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ε, πρόεδρε, σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να συνεχίσουμε τη ζήτηση μας. Ευχαριστώ πολύ Αντώνιο. Συγγνώμη, θα πρέπει να κάνω μια μικρή αλλαγή, αλλά νομίζω πως η κυρία Σουλίνη δεν θα διαφωνεί, διότι ο σκιώδης εισηγητής μας πρέπει να αποχωρήσει, αλλά και ο πρόεδρός μας, Μάλκομ. Γι' αυτό λοιπόν να σου δώσουμε το λόγο πρώτα και μετά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Ελπίζω οι άλλοι σκιώδεις να μην ε, στεναχωρηθούν που θα μιλήσω πρώτος αν θυμόσαστε, είχαμε μία παρόμοια στρατηγική κατά την διαδικασία έγκρισης ε, της οδηγίας ε, μηχανοκίνητων οχημάτων. Ε, βλέπουμε τώρα την ροή των αποφάσεων της Επιτροπολογίας προς την Επιτροπή και είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Πανσέρη θα συμφωνεί ότι είναι μια τυπική διαδικασία. Ε, τώρα βέβαια ως Κοινοβούλιο έχουμε και το δικαίωμα της, του ελέγχου της εποπτείας, ιδίως στον τομέα της επιτροπολογίας και το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την ασφάλεια των μεταφορών, τις, ε, τα, τις ε, εκπομπές καυσερίων κλπ. Όταν είχαμε λοιπόν εγκρίνει τη διαδικασία είχαμε ζητήσει ορισμένες διευκρινήσεις ορισμών και θα ζητήσω το λόγο σύντομα στην Επιτροπή των Περιφερειών να μιλήσω επί του θέματος. Θα πρέπει όμως να συζητήσω προηγουμένως το θέμα με την κυρία Γκέφαρτ για την οδηγία των υπηρεσιών ε, πριν μιλήσω ε, και θα το κάνω αυτό σύντομα για την εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών. Το πρώτο, τώρα για την πρόταση αυτή τη συγκεκριμένη, το πρώτο που ήθελα να πω για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η διαφορά που έχουμε εδώ είναι ότι η Κομισιόν έχει επισημάνει ότι αυτός ο τομέας είναι πολύ πιο ε, ειδικό. Και πολλές μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούν εξειδικευμένα οχήματα όπως ε, σειρώμενα ε, τα οποία διαφέρουν στις προδιαγραφές από τα μηχανοκίνητα οχήματα, από τα αυτοκίνητα. Από την άλλη πλευρά θέλω, χρειάζομαι μια επιβεβαίωση ότι ότι ε, όλα αυτά τα εξαρτήματα ε, απαιτούν ή όχι υποχρεωτική έγκριση. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αναγνώριση των εξαρτημάτων, ιδίως για, το, για τα οχήματα TAF 45 και τα ε, ψηρώμενα εξαρτήματα trailers και γι' αυτό εάν είναι υποχρεωτική η έγκριση για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες τοπικών ελέγχων των εξαρτημάτων αυτών ε, και των, ε, δηλαδή τα 45 και τα ρημουλκούμενα. Εάν αυτό όντως ισχύει θα ε, πρέπει να προσθέσουμε ορισμένες διατάξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το άλλο θέμα, υποχρεωτικό ή όχι λοιπόν, υποχρεωτική ή όχι αναγνώριση. Το άλλο θέμα είναι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών για τα εξαρτήματα των τρακτέρ και αν επιτρέπεται ή όχι να κυκλοφορούν στις δημόσιες οδούς. και τι είδου εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν για να κυκλοφορήσουν στους δημόσιους δρόμους από απόψεως ασφαλείας. Έχουμε κοινά πρότυπα για τρακτέρ τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Το θέμα που πρέπει να διευκολύνουμε η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την πρόσβαση σε αυτήν. Το τρίτο το θέμα στο οποίο υπάρχουν σημαντικές αλλαγές από την Επιτροπή είναι η διάθεση στην αγορά ανταλλακτικών που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις παραμέτρους ασφαλείας των οχημάτων. Όσον αφορά τα μηχανήματα, τα γεωργικά μηχανήματα, ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τι προδιαγραφές ασφαλείας ισχύουν κοίταξα τις προτάσεις και θέλω να εξασφαλίσω ότι η Κομισιόν έχει προσέξει αυτό το θέμα των ε, προτάσεών μας. Δεν βλέπω στην ε, αξιολόγηση επιπτώσεων να αναφέρεται αυτό το θέμα συγκεκριμένα και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για την ε, κοινή, για την κοινή γνώμη δεδομένου ότι έχει επιπτώσεις και περιβαλλοντικές αλλά και επιπτώσεις για τους κατασκευαστές ε, ανταλλακτικών δεδομένου ότι ορισμένοι έχουν δυσκολία πρόσβαση σε αγορές. Επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί από τη μία οδηγία στην άλλη, δηλαδή η πρόσβαση σε τεχνικές ε, πληροφορίες, σε πληροφορίες τεχνικής ε, φύσεως. Όσον αφορά την παλαιότερη οδηγία για τα μηχανοκύματα οχήματα, είχαμε συγκεκριμένε διατάξεις ε, τις οποίες είχαμε εμείς φροντίσει να μπουν στην οδηγία για τις εκπομπές των οχημάτων αυτών και διατάξεις ε, οι οποίες αφορούν την ανταγωνιστικότητα και άλλα στοιχεία των μηχανοκίνητων αυτοκινήτων. Ε, για πολλά χρόνια τα τρακτέρ ε, ανήκαν σε ένα εντελώ διαφορετικό σύστημα, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και όσον αφορά τώρα τις ε, επισκευές, ε, δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι κανόνες και οποιοδήποτε έλεγε ή νόμιζε ότι είχε τις τεχνικές γνώσεις μπορούσε να επισκευάσει τρακτέρ ή γεωργικά οχήματα. Τώρα, από απόψεως πάλι δημόσιας πολιτικής ε, υπάρχουν σαφώς προβλήματα ανταγωνιστικότητας και πρόσβασης σε ε, επιχειρήσεις ε, συντήρησης και επισκευής. Δεν έχει καλυφθεί αυτό το θέμα ότι τη μελέτη επιπτώσεων. Η μελέτη επιπτώσεων δεν αναφέρει αν υπάρχουν επιπτώσεις στο, στη, στο κοινό, στο, στο δημόσιο τομέα διότι εδώ μπλέκουμε με παράγοντες ε, ασφαλείας και με επαγγελματίες, πελάτες. Άλλο είναι η μία μονάδα ε, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και άλλο μία ε, μονάδα επισκευής ε, γεωργικών οχημάτων. Δεν υπάρχει καμία, κανένας περιορισμός ε, πρόσβασης στην εξυπηρέτηση των γεωργικών οχημάτων μέσα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Και γι' αυτό πρέπει να ελέγξουμε αν έχουμε τις κατάλληλες προφορίες στη διάθεσή μας για να ελέγχουμε αυτό τον τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον συγητή να μας στείλει ένα σημείωμα, τον κομισιό να μας στείλει ένα σημείωμα γιατί στη μελέτη επιπτώσεων δεν έχει περιληφθεί αυτό ο τομέας ε, των επισκευαστικών μονάδων ε, για τα γεωργικά αιχήματα και τις επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια. Ε, πιστεύω ότι τότε από την οδηγία αυτοκινήτων είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο αυτό. Υπάρχει στην προηγούμενη οδηγία και θα ήθελα να μεταφαρθεί και σε αυτήν εδώ. Ε, και ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Πανσέρη, για την πολύ ε, εμπεριστατωμένη, λίγαν εμπεριστατωμένη γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Κατρίνη Σιλιέ που είναι η σκιώδης εισηγήτρια. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελέτη επιπτώσεων, η οποία μας διαφώτισε στις νομοθετικές επιλογές που ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με πολύ σαφή τρόπο και υπάρχει και βούληση Επιτροπής να καταλήξει σε απλούστευση κάτι που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Όλοι επιδιώκουμε εναρμόνιση και απλούστευση. Όποτε μπορεί να γίνει, όποτε γίνεται αυτό, πρέπει να το τονίζουμε. Απλούστευση για τι εθνικέ διοικήσει. Εφόσον από το σύστημα τη οδηγία περνάμε στον κανονισμό που περιορίζει το κόστο τη ενσωμάτωση, που είναι σημαντικό, και για τι επιχειρήσει και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μειώνονται ε, τα έξοδα προσαρμογή προσαρμογής ε, στην ισχύουσα νομοθεσία μια, ένα μικρό ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα που έχει επιλεγεί. Πρέπει να ξαναδούμε το νομοθετικό πλαίσιο της έγκρισης τύπου των ελκυστήρων, ενώ μόλις πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ η οδηγία του 2003 τον Ιούλιο 2005 για τα οχήματα νέου τύπου και Ιούλιο 2009 για όλα τα άλλα οχήματα. Μιλάμε λοιπόν για κάτι το πολύ πρόσφατο αν είμαστε αισιόδοξοι μπορούμε να, μιλούμε, μπορούμε να μιλάμε για έξοδο από την κρίση. Αν είμαστε πιο απεσιόδοξοι θα πούμε ότι παραμένουμε σε φάση κρίσης. Οποιασδήποτε τα οικονομικά το οικονομικό βάρος ε, που θα προκύψει από την προσαρμογή ε, ίσως δεν είναι κάτι που θα πρέπει να αναλυφθεί τώρα. Το 2015 όλ, θα πρέπει θα περάσουμε σε νέες φάσεις της οδηγίας για τα καυσαέρια και τη ρήπανση από, μικρο, μικροσωματίδια και πιθανώς να υπάρξει σε μία φάση μία νομική αστάθεια μπορεί λοιπόν να μας επιτρέψει τις επιλογές για ποιο λόγο επέλεξε η Κομισιόν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα. Θα απαντήσει σε λίγο φαντάζομαι η Επιτροπή. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρούλη θέλετε, δεν θέλετε να πάρετε το λόγο. Πολύ ωραία. Ο κύριος Μάντερς ε, ακόμα δεν έχει έρθει. Ο κύριος Φάμπ έχει ζητήσει το λόγο και θα του τον δώσω βεβαίως. Ευχαριστώ. Συγχαίρω την Κομισιόν που επιτέλους μετά από τέσσερα χρόνια που είχε υποσχεθεί ο επίτροπος κύριος Βερχόιγκεν έχουμε αυτή την πρόταση και την έχουμε μελετήσει προσεκτικά. Δεύτερον, μετά από αυτά που, είπε, που είπαν οι δύο ε, εισηγήτριες, δεν ξέρω, σκιώδεις εισηγήτριες, δεν ξέρω κατά πόσον η Κομισιόν έχει χρησιμοποιήσει το άρθρο 44 από την οδηγία των οχημάτων και θα τον χρησιμοποιείται για τους ελκυστήρες για τα τρακτέρ. Διότι το άρθρο 44, αν εφαρμοστεί στα γεωργικά οχήματα, θα πρέπει να ε, αλλάξει σημαντικά, ε, να μεταφερθεί με σημαντικές αλλαγές ε, στη νέα οδηγία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς η Κομισιόν θα μεταφέρει το άρθρο 44 από την οδηγία ε, οχημάτων στην οδηγία για τα γεωργικά οχήματα και συγκεκριμένα για τους ελκυστήρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήπως κάποιος που δεν είναι σκιώδης ηγητής θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κανένας. Κύριε Ματίνο, κύριε Ματίνο, προσπαθώ να το πω σωστά, να το προφέρω σωστά το όνομά σας, δεχθήκατε ε, πολλές ερωτήσεις. Αν μπορείτε να απαντήσετε σε όσο γίνεται περισσότερες ε, ερωτήσεις, θα είμαστε ευγνώμονες. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής για τα εύστοχα σχόλιά τους θα τα λάβω υπόψη μου και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά από αυτά τώρα. Τώρα, αναφορικά με το ζήτημα της προσέγγισης πολλαπλούς επίπεδου και την αναφορά στα διεθνή πρότυπα. Ε, εδώ πρέπει να έχουμε, δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, όχι όλο με βάση την εμπειρία που είχαμε με άλλα ε, οχήματα, αυτοκίνητα, παραδείγματο χάρη πιβατικά αλλά διότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τι ιδιαίτερότητε ε, αυτού του κλάδου των γεωργικών και δασικών οχημάτων. Η, τα διεθνή πρότυπα, τα οποία είναι γνωστά, είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένα. Σε μερικές ε, περιπτώσεις υπάρχουν ε, κάποιες συμβατότητες, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τα σελκυστήρες. Έχουμε πολλά ευρωπαϊκά πρότυπα και ως εκ τούτου η κατάσταση είναι λίγο συγκεχημένη. Αλλά βέβαια νομίζω ότι με την πρόταση αυτή που κάνει προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων και της, της πράξης κατεξοδότηση μπορεί να ε, λαμβάνεται μέσω της επιτροπολογίας ε, με έλεγχο, όπως είπε και ο συγκητής. Μας προσφέρει λοιπόν τα κατάλληλα μέσα για να ασκήσουμε τους απαραίτητους ελέγχους τώρα. Σε ό,τι αφορά Τώρα τα διεθνέ επίπεδο και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην UNEC προτού να εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ ε, χρειάζεται να δοθεί εντολή από τα κρατημέλη προς την Κομισιόν και αυτή η προσέγγιση ε, σχέση με ε, την έλεγχο που ασκείται μέσω της επιτροπολογίας διασφαλίζει παράλληλα και τις ε, απαραίτητες τους απαραίτητους ελέγχους και ισορροπίες προτού να προβούμε στην εφαρμογή αυτών των διεθνών στάνταρ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ισχύοντα πρότυπα, Θα ήθελα να αναφέρω ως παράδειγμα το γεγονός ότι ο κλάδος ε, υπέφερε στο παρελθόν με αλληλεπικάλυψη με άλλα νομοθετήματα και το καλύτερο παράδειγμα είναι η περίπτωση της οδηγίας ε, περί μηχανημάτων. Αναφίβολο ο Σουάμπ θα θυμάται πως ε, τα θεσμικά όργανα, όχι μόνο οι Κομισιόν, ε, έλαβαν θέσεις, κατέβαλαν προσπάθειες μάλλον για να εξορθολογικεύσουν τις, ε, τα πρότυπα αυτά. Και αυτό το πετύχαμε πρόσφατα, το τελευταίο το πετύχαμε πριν από 8 μήνες. Αλλά αναφερόμενοι σε αυτά τα πρότυπα, Απλά λαμβάνουμε υπόψη μας ε, τις καλύτερες ε, τεχνικές ε, προδιαγραφές που μας επιτρέπουν να πετύχουμε τα υψηλά επίπεδα απαιτήσεων που έχουμε θέσει. Να πω επίσης ότι χρειάζεται να εξετάσουμε ποιες είναι οι αναφορές που υπάρχουν στην νομοθεσία περισσότερο στην περίπτωση αυτή που μας απασχολεί τώρα και λιγότερο σε ό,τι αφορά την ε, θέμα αυτοκίνητο αυτοκινητοβιομηχανίας. Τώρα, αναφορικά με το άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τόνισε η κυρία Σούλια θα πρέπει να ακολουθήσουμε προσεκτικά ε, την εκτίμηση αντικτύπου όπου τονίζεται ένα σημείο καμπής ισορροπίας συγγνώμη, για ορισμένα προϊόντα. Μιλήσαμε για κάποια ανταλλακτικά, μιλήσαμε επίσης για κάποια ελκυστήρε που παράγονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τοπική, περιφερειακή ή εθνική αγορά. Και θεωρώ ότι εδώ προστέμενη εδω η προσθεμενη αξια μιας έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκαλεί κάποιο κόστος ελαφρύ μεν, αλλά όπως αναφέρεται και στη μελέτη αντικτύπου, αλλά υψηλότερο με το ισχύον θα επιτρέψει τουλάχιστον να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τον κατασκευαστή να εφαρμόσει την εθνική έγκριση τύπου ή την ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Τώρα να επανέλθω στο ζήτημα που έθιξε ο κύριος Χάρμπουρ το θέμα της ε, αναγνώρισης. Εδώ αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και σε άλλους κλάδους όπως ε, τα ε, βαρικά οχήματα, μοροσυκλέτες κλπ. Η αναγνώριση λοιπόν αυτού του έγκρισης τύπου είναι μια πρόκληση διότι οι απαιτήσει διαφέρουν. Φυσικά οι οριζόντιες διατάξεις ε, της ε, συνθήκης με απαιτήσει ε, κοινοποίηση μπορεί να ισχύουν, αλλά δεν είμαι στη θέση σήμερα να σας επιβεβαιώσω ότι αυτές οι εθνικές εγκρίσεις τύπου θα μπορούν να αναγνωρίζονται και από τις εθνικές αρχές άλλου κράτους μέλους διότι σε μερικέ περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτή η έγκριση αλλά τύπου, αλλά οι απαιτήσει ε, μπορεί να διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Τώρα, η προσέγγιση η οποία επιλέγει στην πρότασή μας ε, είναι αυτή ενός, ε, μιας προσεκτικής προσέγγισης και στόχευσης. Το επιχείρημα του κόστους που άκουσα και ιδιαίτερα το κόστος για τι της επιχειρήσεις. Εάν θέλουμε φυσικά να επεκταθούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα αυτής της αναγνώρισης έγκρισης τύπου, η έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η βέλτιστη των ε, λύσεων. Αλλά για κάποιες ειδικέ κατηγορίες ή υποκατηγορίες αυτή δεν είναι ιδανική λύση, γι' αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο προτείναμε την ε, δυνατότητα επιλογής ε, του κατασκευαστή. Για παντούρα τώρα στο θέμα του συνολικού κόστους του και τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να πω ότι αυτό είναι ακριβώ ο λόγο για τον οποίο και αυτό θα καταστεί σαφέστερο σήμερα το απόγευμα όταν θα μιλήσουμε για τα μοτοποδήλατα και μονομοσυκλέτε είναι ότι εδώ περιορίζουμε τις αλλαγέ σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αλλαγέ σε τεχνικές απαιτήσει το ελάχιστο. Ειδικά επειδή γνωρίζουμε ότι τρέχουσες τεχνικές προδιαγραφές σε ορισμένες πτυχές χρειάζονται οπωσδήποτε ενημέρωση. ενημέρωση ε, επειδή θεωρούνται παγκοσμίω ικανοποιητικά, ικανοποιητικές και ε, λογικές σε κόστος, σε δαπάνες. Ακριβώς λοιπόν αυτό το σκεπτικό απετέλεσε τη βάση των προτάσεών μας για την ελαχιστοποίηση των αλλαγών στην τρέχουσα δέσμη τεχνικών απαιτήσεων. Όσον αφορά αυτή την ε, ε, επικαιροποίηση, τον εξυγχρονισμό των διατάξεων, ε, είναι σε εξέλιξη, ιδιαίτερα στον τομέα της οδικής ασφάλειας και στον τομέα, στον τομέα της πέδησης, των φρεναρίσματος και ε, είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της ε, επικαιροποίησης αυτών των διατάξεων Θέλουμε όμως να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτή την πρόταση και σε άλλες προτάσεις που υιοθετήθηκαν πρόσφατα στον τομέα αυτό. Ε, το έχουμε βάλει κατά μέρο ε, αυτή την πτυχή προς το παρόν, παρόλο που έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση ως μέρος των εφαρμαστικών μέτρων αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Ιδιαίτερα στην πέδηση, ιδιαίτερα σε αυτό τον τομέα υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα για ελκυστήρες με μεγάλες ταχύτητες, για τρακτέρ υψηλών ταχυτήτων. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να το τελειώσουμε αυτό το θέμα πολύ ε, γρήγορα. Είναι έτοιμος ο φάκελος στο σιρτάρι μας αυτό που αφορά δηλαδή τη ρύθμιση όλων των διατάξεων για την πέδηση. Ο στόχος αυτού του είδους της, των νομοθετικών κανόνων είναι, έτοιμος προς, είναι έτοιμα προς έγκριση. Και όσον αφορά τώρα την οδική κυκλοφορία, αυτό εμπίπτει στην ευθύνη των κρατών μελών. Όμως το πλεονέκτημα, το θα είναι ότι θα έχουμε ένα πιο, μια πιο λογική δέσμη διατάξεων και όποτε οι εθνικές υπηρεσίες θα θέλουν να ενημερώσουν, να επικαιροποιήσουν και να εξυγχρονίσουν τις διατάξεις τους, θα μπορούν να το κάνουν αυτό πιο εύκολα. Τώρα θα έχουν ε, οι διατάξεις αυτές μία σημαντική επίπτωση στην οδική κυκλοφορία αυτών του, είδους των μηχανημάτων. Η απάντηση θα είναι, είναι ναι, είναι θετική, όχι άμεσα αλλά έμεσα διότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι προδιαγραφές από τις εθνικές υπηρεσίες όποτε το κρίνουν αναγκαίο από την άλλη πλευρά εναρμονίζουμε ε, τις διατάξεις για τους γεωργικούς και δασικούς ε, ελκυστήρες και ε, πραγματικά εδώ κάνουμε μια εναρμόνιση για αυτά τα οχήματα συνενώνοντας και συντονίζοντας διάφορα κομμάτια νομοθεσίας από εδώ και από εκεί. Τα συγκεράζουμε λοιπόν όλα αυτά σε ένα πλαίσιο εναρμόνισης διότι τότε θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε τα προϊόντα τα οποία ε, συζητούμε σήμερα από την οδηγία μηχανημάτων. Και τέλος, άλλα ειδικά θέματα, το χρονοδιάγραμμα θα το αφήσω τελευταίο. Όσον αφορά τα ανταλλακτικά και τη συντήρηση και επισκευή, για μας ε, τα ανταλλακτικά, η πρόταση αυτή ακολουθεί βασικά την οδηγια 2746. 2007-46 η οδηγία αυτή παρέχει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, την απαραίτητη εξασφάλιση ότι στα ανταλλακτικά έχουμε μία πολύ ικανοποιητική δέσμη προτάσεων. Όσον αφορά τώρα τις επισκευές και τη συντήρηση, καταρχάς ναι, οι διατάξεις δεν αναφέρθηκαν στην μελέτη επιπτώσεων Η μελέτη επιπτώσεων βασίστηκε στις, ε, στα, στα κεκτημένα του 2009 και με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης εξετάσαμε όλες αυτές τις διατάξεις συνεκτικά γνωρίζοντας όμως ότι τα τρακτέρ, οι ελκυστήρες αυτοί δεν είναι ούτε επιβατικά, επιβατικά οχήματα, ούτε μοτοσικλέτες ε, και αυτό που προσπαθούμε να επιφέρουμε με στο θέμα της συντήρησης και επισκευής είναι μία σωστή ισορροπία. Αφενός ε, πρέπει να έχουμε μία ε, έγκριση μία, μία ε, εναρμόνιση των διατάξεων μέσα από διαφορετικές οδηγίες που καλύπτουν ε, διαφορετικούς τύπους οχημάτων και αφετέρου να προσέξουμε τις ειδικότητε του κλάδου. Γνωρίζαμε τις ειδικότητες, τις ιδιαιτερότητες συγγνώμη, του κλάδου αυτού πριν διατυπώσουμε τη μελέτη επιπτώσεων. Και είχαμε συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους ε, του κλάδου εσωτερικά στις υπηρεσίες μας ε, αλλά και ε, με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους και μεταξύ των ενδιαφερομένων του κλάδου όπως είπατε κύριε Χάρμπορ ζητήσατε να τους μεταβιβάσουμε ένα συγκεκριμένο σημείωμα εν ώψη των ε, αλλαγών αυτών για να τους διευκρινίσουμε τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε να επιφέρουμε ε, με αυτή την πρόταση. Κάναμε λοιπόν αυτή τη διαβούλευση πριν έρθουμε εδώ. Όσον αφορά τώρα τη διανομή και τις επισκευές των ελκυστήρων, όλη η διαδικασία δεν είναι ίδια με αυτή των αυτοκινήτων. Έχουμε ιδιαιτερότητες και το ζήτημα είναι ότι τα μηχανήματα ότι αυτά είναι περίπλοκα, όλο και περισσότερα ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά μηχανήματα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται. Επίσης, τις ε, επιχειρήσεις, ε, επισκευαστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα. Έχουμε λοιπόν μία ε, νέα πραγματικότητα από την άλλη πλευρά έχουμε αποκλειστικές αντιπροσωπείες ε, οι οποίες κάνουν τις επισκευές αλλά και τη συντήρηση αλλά και ανεξάρτητες επισκευαστικές μονάδες ε, που αναλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή τρακτέρ. Ε, αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι να μπορούν αυτές οι ανεξάρτητες μονάδες και όλες οι μονάδες συντηρήσεις και επισκευές να έχουν στα χέρια τους τα απαραίτητες πληροφορίες για να γνωρίζουν τις προδιαγραφές που χρειάζονται για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων. Οπότε είμαστε πρόσημοι να διευκρινίσουμε το ερώτημα αυτό με, με ένα σημείωμα το οποίο θα συντάξουμε. και θα ε, περιλάβουμε ε, και την ενημέρωση, θα σας ενημερώσουμε και για τη διαβούλευση που έγινε, διότι αναγνωρίζω ότι δεν σας έχει δοθεί αυτή η ενημέρωση. Για το χρονοδιάγραμμα... Η πρόταση έχει ακολουθήσει ε, δύο διαφορετικά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις η πρώτη ε, προσέγγιση ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε εύλογο χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους του κλάδου να προσαρμοστούν. Αυτό ήταν στη μελέτη επιπτώσεων. Και δεν στοχεύουμε βεβαίως σε τεράστιες αλλαγές ε, τεχνικών προδιαγραφών. Ο στόχος μας δεν είναι να επιβάλλουμε τεράστιες αλλαγές και πιστεύω το χρονοδιάγραμμα είναι επαρκές. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα καυσαέρια. Ο, ο κλάδος των ε, ενδιαφερομένων για τους ελκυστήρες είπε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να παρακολουθήσει ε, τις προτάσεις της Κομισιόν και να υπάρχει ένα ποσοστό ευελιξίας όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τα καυσαέρια, για τις εκπομπές ιδιαίτερα στον ε, ε, δευτερογενή τομέα των μικρών ελκυστήρων, των στενών ελκυστήρων διότι έχουν ιδιαίτερες ε, ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εφαρμοστικά μέτρα και στη κατεξουσιοδότηση πράξης είναι σαφές ότι όταν η πρόταση αυτή την οποία αναλύουμε σήμερα ή αρχίζουμε να αναλύουμε σήμερα, θα αρχίσει να υλοποιείται, να εφαρμόζεται, θα πρέπει να υπάρχουν εφαρμοστικά μέτρα και θα πρέπει οι διάφορες ε, δέσμες εφαρμοστικών μέτρων να είναι έτοιμες. Αυτή είναι μια συνήθις πρόκληση για τις Κομισιόν αλλά και για τα άλλα θεσμικά όργανα. Να ολοκληρώσουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα την ολοκλήρωση της εφαρμοστικής πράξης. μας διευκολύνει το γεγονός ότι εκτός από το τομέα της πέδησης, όπως σας είπα που είναι στο σιρτάρι μας, δεν θα θίξουμε ριζικά τις τεχνικές προδιαγραφές και θα βασιστούμε στην προσέγγιση πολλαπλών επίπεδων, όπως την έχουμε χρησιμοποιήσει και σε άλλες νομοθετικές πράξεις. Είμαστε λοιπόν ε, θετική. Έχουμε, ε, ε, έχουμε λοιπόν μια θετική προσέγγιση και πιστεύω ότι η πρότασή μας είναι επαρκής και σωστή. Ευχαριστώ, κύριε Ματίνο. Το ζήτημα είναι πολύ περίπλοκο, πολύ τεχνικού χαρακτήρα, αλλά είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. το λόγο στον ε, κύριο Μάντερς και μετά θα απαντήσει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> So just, uh, um, no. <laughs> Uh, thank you for... ευχαριστώ που προτείνετε κανονισμό αντί μια ακόμα οδηγία και είναι κρίμα που ο Ανδρέας έφυγε. Α, είναι εδώ, είναι εδώ γιατί ο κανονισμός για έναν τέτοιο τομέα είναι αυτό που απαιτείται και θα έπρεπε να κάνουμε το ίδιο και για άλλους τομείς. Για το θέμα της ασφάλειας θα ήθελα να πω κάτι. Τα γεωργικά και δασικά οχήματα χρησιμοποιούνται συνήθως στην Ήπεθρο, σε στενούς δρόμους. Ε, συνήθως είναι ογκώδη οι ελκυστήρες για να ανταποκρίνονται στις ε, διάφορες ε, ε, στις ανάγκες των αγροτικών εργασιών. Θα ήθελα να πω κάτι για, την άδεια, για το δίπλωμα οδήγησης. Οι οδηγοί είναι 60 ετών και οδηγούν ένα τεράστιο όχημα, μεγαλύτερο από ένα λεωφορείο. Για το να οδηγείς λεωφορείο έχει ειδικό δίπλωμα, ενώ για τα αγροτικά και δασικά οχήματα δεν υπάρχουν καθόλου απαιτήσει. Θα θέλαμε λοιπόν να προβλέψουμε ε, στον κανονισμό την ε, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διπλώματος οδήγησης γιατί μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για συστήματα πέδησης, για αποφυγή ανατροπής. Ε, λοιπόν έχουμε έναν οδηγό που δεν είναι σε θέση να χειριστεί ένα τέτοιο όχημα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Και θα ήθελα να ξέρω αν έχει γίνει κάποια μελέτη για το τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη, για τις άδειε οδήγηση, την ε, ε, ηλικία μετά από την οποία, ποιο είναι το όριο ηλικία για να μπορεί κανείς ε, να οδηγεί, μέχρι πότε μπορεί κανείς να οδηγεί αγροτικά και δασικά οχήματα. Ευχαριστώ. Voilà qui lance. Α, αυτό αρχίζει, αρχίζει, ξεκινάει μια συζήτηση η οποία θα προκαλέσει άλλο στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Αντώνιο για τα συμπεράσματά του τώρα. Sì, Ναι, όντως και αυτό είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται να εξεταστεί διότι το ζήτημα της ασφάλειας ε, είναι ότι δεν ε, κυκλοφορούν μόνο σε αγροτικούς, αγροτικές περιοχές και σε αγροτικούς δρόμους, αλλά για να μετακινηθούν πρέπει να διασχίσουν και κάποιους δρόμους οι οποίοι είναι πολύ σύχναστοι κλπ. Λοιπόν, να πω ότι συνεχίζω να έχω κάποιες αμφιβολίες αναφορικά με το ζήτημα της επιλογής εθνικής, ε, εθνικός τύπος έγκρισης ή ευρωπαϊκός ε, τύπος πως ε, μερικές φορές υπάρχει κίνδυνος ε, να βρεθούμε σε σύγκρουση με τα όσα φτιάχνουμε εμείς στην Ευρώπη και τα όσα γίνονται στην ε, ακράτη μελη και το ζήτημα των ανταλλακτικών επίσης είναι ένα θέμα καυτό. Το εμβαθύναμε όταν ασχοληθήκαμε με την έγκριση των μηχανοκινήτων οχημάτων. Νομίζω ότι κατά τα υπόλοιπα υπάρχουν περιθώρια για να κάνουμε μια αποτελεσματική δουλειά και μια αποτελεσματική συνεργασία. Ευχαριστώ για την Κομισιόν για τη συνεισφορά τη. Ευχαριστώ Αντώνη. Θα σας ε, αναφέρω τώρα το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε. Α, είναι προσωρινό. Είναι προσωρινό. Θέλετε το πρώτο χρονοδιάγραμμα, όχι. Τότε περνάμε στο επόμενο σημείο. Το οποίο όμως είναι εντελώ διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η συνέχεια των εργασιών μας ε, που ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια. Περνάμε στην οδηγία περί υπηρεσιών και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια Εύλεν Γκέμπαρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που μόλις είπατε. Η οδηγία υπηρεσιών θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια πολλές φορές. Διότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά νομοθετικά κείμενα και σε τέτοια περίπτωση όχι μόνο νομοθετούμε αλλά θέλουμε να εποπτεύσουμε και την εφαρμογή και ε, την εφαρμογή των διατάξεων και να έχουμε και την εποπτεία, την παρακολούθηση των εξελίξεων για να δούμε ε, ε, την πρόοδο και έχουμε επίσης υποβάλει ορισμένες, ε, ε, ορισμένα ερωτήματα στην ε, Επιτροπή, στην Κομισιό όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας. Δεν προσπάθησα να... δεν ήμουν πολύ φιλόδοξη σε αυτή τη γνωμοδότηση γιατί δεν πρέπει να έχουμε μεγάλες ε, προσδοκίες διότι πολλές, πολλά κράτη-μέλη μετέφεραν την οδηγία πάρα πολύ αργά, υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις και έτσι ήταν πολύ δύσκολο να έχω μία γενική εικόνα. Παραδείγματο χάρη, με ρώτησαν και οι δημοσιογράφοι ε, πολλές φορές κάποιο κινητό, ακούγεται, ο κύριος Σβάμπ τρέχει να το πιάσει. Ε, <laughs> έχουμε λοιπόν όχληση από το κινητό και μουσική ε, ευχάριστη. Κάποιο μωρό, το κινητό έχει έναν ήχο ε, μωρού που φώναζε, που έκλαιγε. ευχάριστη διακοπή ήταν αυτή, λέει η κυρία Γκέπαρτ. Ακούσαμε λοιπόν το μωρό αλλά εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με τα δικά μας. Λοιπόν, με ρώτηση σαν δημοσιογράφοι, ε, Πόσε θέσει απασχόληση δημιουργήθηκαν με την οδηγία αυτή. Ε, δεν μπορώ να απαντήσω σε ένα τέτοιο ερώτημα, δεν είναι καθόλου απλή απάντηση. Και επίσης η μεταφορά της οδηγίας αυτής, αυτό μελέτησα εγώ στα κράτη-μέλη, όχι την, τις επιπτώσεις, αυτό θα γίνει αργότερα όταν θα έχουμε και την πρώτη έκθεση της Κομισιόν, την πρώτη την ε, περιμένουμε την άνοιξη του χρόνου. Σύμφωνα με αυτά που, που είχαμε πει, ε, ε, πρόσεξα τέσσερα σημεία ιδιαίτερα και η έκθεση επικεντρώνεται σε αυτά. Ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές που μου έδωσαν τις ε, παρατηρήσεις τους, μου υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους εγκαίρως για να μπορέσω να τις ε, μελετήσω για την ε, σύνταξη της έκθεσης. Ιδιαίτερα πάλι σε θέματα μεταφοράς της οδηγίας υπηρεσιών. Βάσει αυτών που συμφωνήσαμε, ζητάμε μια αξιολόγηση της οδηγίας για να δούμε πώς μεταφέρθηκε στα κράτη-μέλη το screening. Στην οδηγία υπηρεσιών ε, ε, είπαμε ότι στο κράτος μέλος όπου οι διατάξεις πρέπει να, πρέπει να γίνουν σεβαστές πρέπει επίσης να εξετάσουμε ακριβέστατα εάν οι κανόνες ε, που ισχύουν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ε, της εσωτερικής αγοράς και δεν, είναι ε, δεν συμβάλλουν στον προστατευτισμό. Τα αφενός λοιπόν σεβασμό των διατάξεων αφετέρου προσοχή στον μη τυχόν υπάρχουν προστατευτικές πτυχές προστατευτισμού. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ανέλαβαν τη δέσμευση να εκτελέσουν μία αμοιβαία αξιολόγηση. Ε, σήμερα στην πολιτική συζήτηση ε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ήμουν τότε προβουλευτής και μου είχαν πει τότε τα, τα κράτη-μέλη αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτή η αμοιβαία αναγνώριση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Εν συνεχεία υποβάλαμε την πρόταση στην Κομισιόν η οποία διέγραψε ένα τμήμα της πρότασής μου ενώ οι υπουργοί το ξανάβαλαν μέσα στην πρόταση. Σήμερα η κατάσταση είναι αντίστροφη. Έχω αλλάξει προσέγγιση και ο κύριος Σβάμπ έχει αλλάξει τη γνώμη του διότι πιστεύουμε ότι η αμοιβαία αναγνώριση μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο μέσο για να παρακολουθήσουμε τι έχει γίνει, πώς εξελίσσεται η εφαρμογή της οδηγίας και επίσης μπορεί να επιβάλλει περισσότερη διαφάνεια. Σημαντικό λοιπόν εργαλείο, σημαντικό μέσο. Θα, δεν θέλω να διαβάσω, να σας διαβάσω μερικές παραγράφους, αλλά, ορισμένες παραγράφους, αλλά ε, επανερχόμεθα συνέχεια σε, ένα, σε μερικά σημαντικά σημεία ε, Αναγνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών ε, ε, προσόντων και, και διπλωμάτων. Αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία ε, στην εσωτερική αγορά. Και ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες παραδείγματος χάρη. Έχουμε συζητήσει τέτοιες ιδέες και άλλες οι οποίες δεν περιέχονται στην ε, οδηγία υπηρεσιών. Είχαμε συμφωνήσει ότι τέτοιου είδους ε, ζητήματα δεν θα καλυφθούν. Έχουν όμως επιπτώσεις στην εφαρμογή και στη μεταφορά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Όλη η διαδικασία της αξιολόγησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Από τη μία πλευρά συνεπάγεται διοικητικών ε, ενεργειών, ε, από την άλλη πλευρά υπάρχουν και πολιτικές πτυχές. Εγώ πιστεύω ότι το, η πολιτική πτυχή έχει περισσότερο βάρος, ε, διότι η όλη οδηγία έχει πολιτικό περιεχόμενο και μας ενδιαφέρει να δούμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν δίκαια και ισότιμα στην ε, εφαρμογή των διατάξεων, παραδείγματος χάρη στο θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Και είναι κρίμα που δεν, δεν έχουν προχωρήσει τα κράτη-μέλη σημαντικά και ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Δεύτερον, Δεύτερον, έχουμε τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Εδώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σκέλος στην οδηγία υπηρεσιών, διότι εδώ θα μπορούμε να βοηθήσουμε με τα κέντρα αυτά σημαντικά τους ε, εξυπηρετούμενους, τους ε, πελάτες, τους ενδιαφερόμενους παρόλο που υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά τη διαμόρφωσή τους. Πρέπει να πω ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει πολύ ικανοποιητικά για τη διαμόρφωση αυτών των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης όπου τα οποία κέντρα μπορούν και διανύμουν ε, πάρα πολλές ε, πληροφορίες και βοηθούν τους ενδιαφερόμενους σε διάφορα στις αιτήσει τους, ε, όχι μόνο στην ενημέρωση αλλά και πρακτικά. Άλλα κράτη-μέλη είναι πιο επιφυλακτικά όσον αφορά τις υπηρεσίες των κέντρων αυτών και είναι περισσότερο κέντρα ενημέρωση. Λειτουργούν περισσότερο ως κέντρα πληροφόρησης. Υπάρχουν επίσης κράτη-μέλη τα οποία είχαν πολλά τέτοια κέντρα εξυπηρέτησης και άλλα ελάχιστα. Ε, σε ορισμένα κέντρα εξυπηρέτησης διευκολύνεται η ζωή των ε, ε, πολιτών, σε άλλα όχι. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτά τα κέντρα εξυπηρέτησης πώς λειτουργούν και ενδεχομένως να βελτιώσουμε την λειτουργία τους εκεί όπου χρειάζεται. Επίσης, σε ποιες γλώσσες το γλωσσικό ζήτημα. Ε, σε ποιες γλώσσες θα προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες. Εδώ ο κύριος Λόγκαρντ έχει και η κυρία Χάνσλικ είχαν ορισμένες παρατηρήσεις σημαντικές τις οποίες έλαβα υπόψη. Θα, καταρχάς μιλούμε για την γλώσσα του κράτους μέλους αυτό είναι βεβαίω ε, λογικό. Όμω, καλό θα ήταν να παρέχονται υπηρεσίε αυτέ και σε άλλε γλώσσε. Παραδείγματο χάρη στη γλώσσα των κρατών που συνορεύουν ε, με το κράτος της έδρας του κέντρου, παραδείγματο χάρη στα πολωνικά στη Γερμανία, όπου έχουμε μεγάλα σύνορα. Ε, έτσι ώστε να υπάρχει λοιπόν και διασυνοριακή γλωσσική εξυπηρέτηση. Πιστεύω ότι εάν ένας ε, Φινλανδός θέλει να εργαστεί στην Ελλάδα, καλό θα ήταν να προσφέρονται οι πληροφορίες και εξυπηρέτηση σε μια άλλη γλώσσα πλην των ελληνικών, τουλάχιστον σε μια άλλη γλώσσα. Και ε, επίσης λυπάμαι που τότε, ε, οι πρώτες που είχα κάνει παλιότερα, να οργανώσουμε ένα συντονιστικό κέντρο ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είχε τύχη της πλειοψηφίας και η Κομισιόν δεν είχε υποστηρίξει, δεν είχε δει θετικά την πρότασή μου αυτή για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κέντρο Ίσως στα πλαίσια τώρα της έκθεσης θα μπορούσε η Κομισιόν να ξαναμελετήσει την πρόταση αυτή και να δει ποια μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ποια κέντρα μπορούμε να οργανώσουμε έτσι ώστε να υπάρχει πανευρωπαϊκή πρόσβαση και εξυπηρέτηση. Äh, Ιδίω για κράτη-μέλη όπου όλο το θέμα αυτό έχει καθυστερήσει πολύ. Εν συνεχεία, διοικητική συνεργασία. Εδώ το θέμα της συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική διότι έχουμε πολλές αρμοδιότητες, διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται πρέπει να εξασφαλίσουμε έναν αποτελεσματικό έλεγχο του, του, του, του, του υπηρεσιών στον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια και, το, και επίσης να χρησιμοποιηθεί το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς, το ΙΜΗ. Αυτό πρέπει να διευρυνθεί και να εδρεωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Ε, ε, και έτσι ώστε οι υπάλληλοι στα κράτη-μέλη να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ικανοποιητικά ε, τους πολίτες. Και τέταρτον και τελευταίος τομέα στον οποίο αναφέρουμε είναι το πεδίο εφαρμογής. Σε ορισμένα κράτη-μέλη έγιναν συζητήσεις με εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών. Παραδείγματο χάρη. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα. Στη Γαλλία, στη Γαλλία πώς θα γίνει η διαχείριση του αποκλεισμού των εξαιρέσεων ορισμένων τομέων των υπηρεσιών, διότι είχαμε πει ότι ορισμένοι τομείς μπορούν να εξαιρεθούν βάσει αποφάσεων των εθνικών αρχών. Αυτή ας πούμε η συζήτηση έγινε στη Γαλλία, γίνεται και στην Πολωνία. Παραδείγματο χάρη, οι Πολωνίοι μα ζητούν. Δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερου τομεί στι υπηρεσίε. Το ένα κράτος θέλει εξαιρέσεις, το άλλο κράτος θέλει αύξηση των τομέων που περιλαμβάνονται. Ε, έχουμε λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εδώ μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια οδηγία η οποία προσπαθεί να οριστικοποιήσει το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών ε, έτσι ώστε να καλύπτονται αυτά τα οποία εμείς έχουμε ορίσει στο ελάχιστο επίπεδο και εν συνεχεία αφήνεται στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών αυτά τα οποία μπορούν να ρυθμίσουν μόνοι τους. Είχα χρονική πίεση, χρονικό περιορισμό για την υποβολή της εξαίσεως ε, δεν έχω υποβάλει ακόμα τις τροπολογίες, δεν τις έχετε, αλλά οπωσδήποτε θα τις παρουσιάσω και θα υποβάλω θα, θα σας παρουσιάσω τις τροπολογίες. Υπάρχει ένα ζήτημα που στην τελευταία συνεδρίαση που είχαμε κάνει με τους οι εισηγητές, ένα ζήτημα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν θα πρέπει να το περιλάβω ή όχι. Εγώ θα ήθελα να περιλάβω αυτό το ζήτημα. Αλλά θέλω να έχω τη συμφωνία σας. Στην οδηγία υπηρεσιών, ό,τι έχει να κάνει με το φορολογικό καθεστώς, όλα αυτά έχουν εξαιρεθεί. Δημοσιονομικές φορολογικές πτυχές έχουν εξαιρεθεί. Όμως, όπως διαπιστώσαμε στις συζητήσεις μας και με τους κοιόδης, αλλά και με άλλους, με άλλα άτομα που εργάζονται στον τομέα αυτό μου, μας είπαν ότι τα κέντρα αυτά δεν σας διαθέτουν πληροφορίες για τον ΦΠΑ, για το καθεστώς φορολόγησης, για το καθεστώς ε, ασφάλισης αυτό το ας πούμε παράπονο το έχω ακούσει από πολλούς ενδιαφερόμενους διαφόρων κλάδων που μου λένε νομίζουμε ότι είναι λογικό αυτού του είδους οι πληροφορίες οικονομικής φύσης περισσότερο να παρέχονται επίσης. Θέλω λοιπόν, θα ήθελα να συμπεριλάβω και αυτό το ζήτημα εκφράζοντας μία παράκληση στην Κομισιόν να εξετάσει πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτό το αίτημα. Παραδείγματο χάρη όταν ένας εργαζόμενος ε, ε, λάβει πληροφορίες για το πώς θα πρέπει να εργαστεί, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, αλλά καμία πληροφορία για τη δικαιώματά του, ούτε για το πώς θα φορολογηθεί, πώς θα καλύψει τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, τι δικαιώματα έχει κλπ είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Τι ΦΠΑ θα πληρώσει, αν θα πληρώσει κλπ. Ε, είναι μία, ένα κενό αυτό. Είναι μία ε, έλλειψη η οποία σημειώνεται σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως είναι επίμαχο το θέμα, γι' αυτό και εξαιρέθηκε. Επειδή θέλαμε να αποφύγουμε τους, τους Αυτό λοιπόν ήθελα να ζητήσω και ολοκληρώνοντας σε όλη τη συζήτηση ε, που έχουμε ε, θα σήξουμε το θέμα του φορολογικού, της φορολογικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αρχίσω όμως τη συζήτηση αυτή σήμερα, αλλά απλώς σας ε, παρουσιάζω την προοπτική του μέλλοντος. Δεν θα αποφύγουμε αυτό το θέμα και αφήνω το λόγο στους κοιόδους ηγητές προς το παρόν. Ευχαριστώ Ευλίν. Νομίζω ότι στο τέλος της παρέμβασής σου έθεσες πολύ θεμελιώδη ερωτήματα και εφόσον έχει έρθει η Επιτροπή και χαιρετώ, το τα, τους εκπροσώπους της ε, διότι με την κρίση έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οτροπία. Ε, και αυτό είναι ίσως ένα θετικό στοιχείο, ίσως είναι ένα θετικό στοιχείο αυτό, το μόνο θετικό στοιχείο της κρίσης. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Άτσλικ, η οποία εκπροσωπεί το ΕΛΚ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία εισηγητή για μια πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική έκθεση. Για μένα υπογραμμίζει τα πιο σημαντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Έχω μόνο ένα σχόλιο κριτικής που αναφέρεται στο σημείο 18. Το είχαμε συζητήσει όταν συναντηθήκαμε με τους σιώδεις εισηγητές. Λέτε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν δυσκολίες να προσδιοριστούν οι εξαιρεσει όταν μιλάμε για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες ειδικότερα. Δεν έχω όμως βρει οποιαδήποτε επιβεβαίωση αυτού του, αυτής της δήλωσης, αυτής της διαπίστωσης ήρθα σε επαφή με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, μελέτης, εξέτασα μια μελέτη που είχε αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι μια δήλωση που με προβληματίζει και σχετίζεται με τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ και θα έρθει και σε εμά όταν θα μιλήσουμε για το μέλλον των υπηρεσιών ε, δημοσίου και γενικού συμφέροντος. Θα έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τα άλλα σημεία αυτού του κειμένου δεν έχω καμία κριτική παρατήρηση να κάνω. Όπως είπα προηγουμένως, κάνατε θαυμάσια δουλειά. Θα ήθελα να διευρυνθεί η έκθεση σε τέσσερις τομείς. Στο κείμενο, στο κείμενο είδα μια αναφορά στο σύστημα εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων ή αδειών ενώ σε άλλα σημεία δεν είχαν διαγραφεί καθόλου. Μα θυμίζει επίση, η κυρία ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το δικό του σύστημα και τις δικές τους απαιτήσει, κάτι που δεν το αμφισβητώ, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η αναθεώρηση αυτού του συστήματος αδειοδότησης έχει ουσιαστικά οδηγήσει στην κατάργηση, την τροποποίηση των συστημάτων οι οποίοι ε, δεν έχουν, δεν έχουν αναλογικότητα ή μπορεί να καταλήξουν σε διακριτική μεταχείριση. Αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει κάπως και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε σχετικά με αυτό το θέμα. Κάτι που θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ίσως περισσότερο είναι ότι αυτά τα, τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης θα πρέπει να ενισχυθούν, να προβάλλονται όλο και περισσότερο και να βελτιώνονται από τα κράτη-μέλη, όχι απλά να ιδρυθούν και μετά να μην γίνει καμία προσπάθεια για την ε, διεύρυνση των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. Έτσι όπως τα περιγράφετε, φαίνεται ότι θα είναι φιλικά προς τους ε, χρήστες και οπωσδήποτε θα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα είναι χρήσιμα για τους χρήστες. Διοικητική συνεργασία. Χωρίς διοικητική συνεργασία δεν μπορεί να λειτουργήσει η οδηγία. Αλλά κατά την άποψή μου η οδηγία αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται ε, ε, ε, μεταξύ πρέπει να, εφαρμοστεί σε συνεργασία όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Αρχές αλλά και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Διότι μόνο τότε θα, είναι, θα στεφθεί με, πραγματικά με επιτυχία η όλη διαδικασία. Μιλήσατε για την αξιολόγηση από ομότιμους Είπατε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να γίνει αξιολόγηση του συστήματος. Αυτή η αξιολόγηση, η αμοιβή αξιολόγηση, η αξιολόγηση από ομότιμους θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω βάρος για τις διοικητικές υπηρεσίες. Πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έχω μιλήσει με εκπροσώπους της διοίκησης στην Πολωνία και αυτό που άκουσα είναι ότι ήταν πολύ σημαντική πρόκληση να προβούν οι ίδιοι οι υπάλληλοι της ε, διοίκησης στην αξιολόγηση η οποία οδήγησε σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Μου είπαν επίσης ότι έκαναν αυτή την άσκηση, έτσι τη χαρακτήρισαν. Και όταν έλαβαν μέρος στην αξιολόγηση, την αμοιβαία αξιολόγηση, την αξιολόγηση από ομότιμους, τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν τι συνέβαινε στις άλλες χώρες. Διδάχθηκαν από αυτή την ανταλλαγή και είναι λοιπόν μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ κρατών μελών. Και κάτι που ασφαλώς θα συζητηθεί στο μέλλον είναι το φορολογικό και το δημοσιονομικό θέμα, το οποίο το αφήνω επί του παρόντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση μιας μελέτης για να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες των κρατών μελών. Πάντως, ε, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, έκανε θαυμάσια δουλειά και ε, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία για περαιτέρω εργασίες. Τώρα ερχόμαστε στον σκιώδη συγητή. Τον κύριο Λούκινγκάρτ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκέμπαρτ για την επικοδομητική συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας. Οι παρατηρήσεις μου ε, συμπεριλήφθηκαν στην έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Όπως είπα και την περσμένη εβδομάδα, πρόκειται για μια πολύ καλή και πολύ ισορροπημένη έκθεση στοχεύει στην εφαρμογή και όχι στα προδοσιακά επίμαχα ζητήματα του παρελθόντος. Αυτό είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Ο... Για Γκέμπαρντ ακόμα δεν έχουμε μια πλήρη εφαρμογή της ε, οδηγίας περί υπηρεσιών όπως δηλώνετε κι εσείς. Ε, αυτό είναι αποδεκτό. 16 κράτη-μέλη εφαρμόζουν την οδηγία και 5 δεν έχουν ε, ακόμα προχωρήσει στα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να προχωρήσει τώρα η οδηγία αυτή. Τώρα αναφερθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο αφορά το κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης. Χρειάζεται να τονίσουμε περαιτέρω το γλωσσικό ζήτημα Χαίρομαι που το λαμβάνετε και εσείς υπόψη σας τα σοβαρά και το τονίζετε στην έκθεσή σας. Κάτι ακόμα για το θέμα της ε, των ε, κέντρων εξυπηρέτησης τα οποία θα πρέπει να φιλικά προς τον χρήστη είναι δύσκολο σήμερα όταν μιλάμε για ηλεκτρονικές ε, υπογραφές αν όχι αδύνατον να εφαρμοστεί σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό εφαρμόζεται περισσότερο σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό φυσικά αποτελεί ένα πρόβλημα για τους αλλοδαπούς που εργάζονται σε μια άλλη χώρα. Στην Ιταλία άκουσα ότι ε, κάποιος που δουλεύει θα πρέπει να μεταβεί στη Ρώμη για να πετύχει αυτή την ηλεκτρονική υπογραφή και μετά να επιστρέψει στην πόλη στην οποία εργάζεται. Τώρα, ηλεκτρονικές υπογραφές δεν πρέπει να απαιτούνται από όλους τους παραγωγούς υπηρεσιών από τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης. Αυτό συμβαίνει σε μερικά κράτη. Σύμφωνα με την οδηγία ξέρω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν μια αξιολόγηση αντικτύπου αναφορικά με το πότε απαιτείται αυτή η ηλεκτρονική υπογραφή. Χρειάζεται να τονιστεί περαιτέρω λοιπόν στην έκθεση σας. Και μια ερώτηση, δεν ξέρω αν θα ήταν δυνατόν, αλλά θεωρώ ότι είναι λογικό να ζητάμε για μία ενιαία ηλεκτρονική υπογραφή για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Το θέτω το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν εφικτό να γίνει κάτι να όψει μου και αυτό θα επέλει πολλά από τα ζητήματα που προανέφερα. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν αυτό το ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής υπογραφής. Ερωτηματικό. Όπως είπε η κυρία Γκέπαρτ, το θέμα των ε, των καθηκόντων πώς θα λειτουργούν λοιπόν αυτά τα κέντρα. Π.χ. το ζήτημα του ΦΠΑ. Νομίζω ότι Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τώρα, για τα κέντρα ενίσχυση εξυπηρέτηση και την αμοιβαία συνεργασία αυτών των κέντρων. Χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά τα κέντρα. Και κάτι τελευταίο σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, η περίφημη παράγραφος 18 όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα. Δεν ε, έχω καταλάβει απόλυτα περί τόνος πρόκειται και ε, ήθελα να ζητήσω από την κυρία Γκέμπερτ αν θα μπορούσε να με διαφωτίσει περί αυτού. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κόφλαν, σκιώδη συγκητής για την ομάδα των Πρασίνων. Καλημέρα σας. Θα απευθυνθώ απευθείας ε, στην Ευλίν και στους σκιώδεις εισηγητές που ε, ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είχαμε ήδη μια συνεδρία εργασίας για αυτό το θέμα. Ε, σημείωσα, έλαβα γνώση αυτών που είπατε τότε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο για να καταλήξουμε στις συμβαστικές λύσεις. Διαβάζοντας την έκθεση, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που είναι το πλαίσιο της πράξης για την ενιαία αγορά που λέει αφενός ότι η δημιουργία της ενιαίας αγοράς, θα οδηγήσει σε τέσσερα σημεία ανάπτυξη όπω λέει ο Μισελ Μπαρνιέ. Ακούσαμε πάρα πολλά στοιχεία αριθμητικά στην οδηγία για τις ε, υπηρεσίε ότι θα δημιουργήσει θέσει εργασία, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ νωρί να το κρίνουμε αυτό ή να πούμε το αντίθετο αλλά και πάρα πολύ νωρί για να ξεκινήσουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Ότι φυσικά επειδή θα το κάνουμε αυτό θα δημιουργήσει θέσει εργασία, θα ε, ε, στηρίξει την ανάπτυξη αλλά δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Υπάρχει και το μακροοικονομικό πλαίσιο που πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη. Θα είχα λοιπόν την τάση να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που έχουμε στο τραπέζι, όπως συνέβη και ε, για την οδηγία για τις υπηρεσίες σχετικά με την ε, πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με το Single Market Act λέγεται σε, στο, κείμενο, ορίζεται σε, αναφέρεται στο κείμενο ότι ο τρόπος που εφαρμόστηκε η οδηγία των υπηρεσιών έχει δώσει κάποια στοιχεία και κάποιες αποδείξεις. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την πρόταση διότι ακριβώς εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ε, στο οποίο λέει ότι έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οδηγία αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι νωρίς να λέμε ότι αυτή είναι η ικανοποιητική και κατάλληλη μέθοδος. Γι' αυτό θα ήθελα να ενισχύσω το στοιχείο της αξιολόγησης και της αποστασιοποίησης που προβλέψατε εσείς. Τώρα, για την ε, οδηγία ε, σχετικά με την υπηρεσία δημόσιου συμφέροντος. Δεν είναι η στιγμή να ξαναρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν τεχνικοί και πολιτικοί λόγοι για τους οποίους δεν είναι σκόπιμο να κάνουμε κάτι τέτοιο, ε, λαμβάνοντα υπόψη τι δυνητικέ πλειοψηφίε στο Κοινοβούλιο. Παράλληλα όμω, μετά τη, όταν θα μιλήσουμε για το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, την υπηρεσία δημόσιου συμφέροντος, επειδή αυτό το κείμενο ε, θα αποτελέσει αντικείμενο σοβαρή συζήτηση με την Βελγική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες που μας προσφέρει φέρει η συνθήκη της Λισαβόνας και στον σκόπο να προσθέσουμε μια πρόταση η οποία θα καλεί, θα ζητά την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι με εντυπωσίασε αυτό που είπατε για τα δικαίωμα σε εργασία, το, την ενημέρωση για, το φορολογικό καθεστώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που παρέχονται, ενώ στο, κάτι που δεν είχα βρει στη γραπτή ε, έκδοση, ε, του, εκδοχή του κειμένου. Και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε χώρο στο κείμενο για αυτό το πολύ σημαντικό που είπατε έστω και να, αυτό σημαίνει να περιορίσουμε αυτά που λέμε για τα κέντρα νέας εξυπηρέτησης ε, για να προσθέσουμε μία παράγραφο που θα περιλαμβάνει αυτά που είπατε και που θεωρώ πάρα πολύ σωστά. Θα απαντήσει η Εύλην σε λίγο. Επειδή θα χρειαστεί να φύγω, να σας εγκαταλείψω, θα αφήσω τη θέση μου στη συνάδελφο. Επειδή δεν θα έχω τη δυνατότητα να μιλήσω λοιπόν εφόσον θα φύγω, θέλω να πω και εγώ ότι συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνουμε απολογισμό. Ε, διότι από αυτό εξαρτάται η αξιοπιστία τόσο της ε, Επιτροπής όσο και του Κοινοβουλίου. Μήπως θα θέλετε να μιλήσετε εξ τη κυρία Σουένσον που δεν είναι παρούσα. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Όχι. Πολύ ωραία. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μάντερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Εύελιν, διότι είναι πραγματικά απόλυτα ισορροπημένη η εκθεσή της. Διότι όταν πριν μερικά χρόνια συζητήσαμε το θέμα, υπήρξε μια συναισθηματική, θα λέγαμε, φόρτιση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, αλλά όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο Όλοι φοβούμασταν τότε το μέλλον. Φοβούμασταν τον ε, Πολωνό Ιδραυλικό. Αλλά τελικά τίποτα δεν συνέβη. Ακόμα και οι Γάλλοι, ο Γάλλος συγγνώμη, πρέσβης παρουσίασε μια έκθεση νομίζω πως ε, η ε, αξιολόγηση από τα κράτη-μέλη ανακλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στις χώρες τους. Ο Γάλλος ε, πρέσβης λοιπόν ήταν απόλυτα ευχαριστημένος ε, από το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης διότι θεώρησε ότι θα μας απαλλάξει από ένα διοικητικό άχθος. Ε. Σήμερα κοιτάζουμε πώς έχει εξελιχθεί το ζήτημα και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί όμως ένα άχθος ακόμα και για τους Γάλλους παρόχους. Εντάξει, μολονότι ήταν ιδιαίτερα θετικό λοιπόν ο πρέσβη τότε για την οδηγία περιπηρεσιών. Σα ευχαριστώ λοιπόν κυρία Γκέμπαρτ. Του λεχθέντο να πω ότι επειδή άκουσα κάποιες ιδέες αναφορικά με κάποιες πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα, φορολογικού κλπ. Αυτό ναι, φυσικά έχει σημασία για αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν και να εργαστούν σε άλλη χώρα. Φυσικά η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική υπογραφή θα πρέπει να καταστεί δυνατή, διότι όπως είπαμε βρισκόμαστε στην ενιαία αγορά και θα πρέπει να πάμε και ακόμα παραπέρα και να πούμε ότι θα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος αριθμός ΦΠΑ δεν θα πρέπει λοιπόν να προσφεύγεται στα εθνικά συστήματα λόγω του ΦΠΑ, διότι ο ΦΠΑ είναι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και κάτι ακόμα, δεν θέλω να δείξω όμω εδώ το κουτί τη Πανδώρα, αλλά ίσω τώρα βρισκόμαστε σε κάπω πιο ήρεμα νερά από ό,τι στο παρελθόν. Βρισκόμαστε λοιπόν στο μέλλον της συζητήσεως που είχαμε στο παρελθόν. Ίσως ε, θα πρέπει να άρουμε κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες ε, παρεκκλήσεις. Ε. Να αναρωτηθούμε λοιπόν ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να αποκλείονται, να εξαιρούνται. Αυτό θα μπορούσαμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε και να άρουμε κάποιες από τις εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρμογή ίσως να χρειαστεί να εξετάσουμε τι, ε, ποιες εξαιρέσεις ε, μπορούμε να άρουμε διότι δεν θα πρέπει πλέον να φοβούμεθα ότι μας ε, ότι απειλούν, απειλούν τα εθνικά μας συστήματα. Ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να το σκεφτούμε το ζήτημα και νομίζω ότι η πρόταση είναι καλή. Ευχαριστώ. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου. Ο κύριος Μάντελς ε, ε, αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα το οποίο είναι κάπως ολιστηρό, παρακινδυνευμένο να ξανανοίξουμε. Θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο και ε, κυρία Γκέμπαρτ. Ναι, ναι, πολύ γρήγορα. Δεν θα υποστηρίξω την τρελή ιδέα του κυρίου Μάντερς. Η βασική μας επίκριση ήταν ότι δεν γίνεται διαφορά μεταξύ της ε, παροχής υπηρεσιών επαγγελματικών και υπηρεσιών του δημοσίου. Γι' αυτό ακριβώς ε, υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Πάντως δεν θα ακολουθούσε την δική του ιδέα. εγώ ενδιαφέρομαι για το screening. Στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή και εδώ όταν ο κύριος Μπανιέ ήταν μαζί μας είχαμε συζητήσει για το screening και στη μεταφορά της οδηγίας ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα. Στη Γερμανία π.χ. το screening γίνεται υπερβολικά λεπτομερός. Κάθε 12.000 κοινότητες, ανά 12.000 Ζητείται υπαρχή πληροφοριών για το πώς ε, ε, διαχειρίζονται τα νεκροταφεία τους, πόσες λάμπες ε, στους δημόσιους δρόμους έχουν φωτισμού. Λοιπόν, δημιουργείται περισσότερη γραφειοκρατία και όχι απλούστευση, ιδίως σε τομείς που είναι εντελώς άσχετοι για την εσωτερική αγορά διότι η εσωτερική αγορά δεν ενδιαφέρεται ούτε για πόσα φώτα καίει μία κοινότητα, ούτε για πόσες, ε, ε, σε, σε τι διάστημα υπάρχει μεταξύ των τάφων σε ένα νεκροταφείο. Λοιπόν, να επικεντρωθούμε στην ε, ουσία και να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ κύριε Ρίλε. Και τώρα το λόγο στην Κομισιόν, η κυρία Μαρτίν Πράτ. Ευχαριστώ. Καταρχάς ήθελα όπως οι σκιώδεις εισηγητές να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της η οποία αναγνωρίζει τη σημασία της οδηγίας υπηρεσιών και η έκθεσή της είναι πολύ επικοδομητική προσπαθώντας να συγκεράσει τις ε, διάφορες ομάδες και τις διάφορες πτυχές από εδώ και από εκεί για ένα θέμα το οποίο είναι λίγα σημαντικό για την εσωτερική αγορά. Θα προσπαθήσω στις διάφορες ερωτήσεις που τέθηκαν ε, και στις παρατηρήσεις. Καταρχάς, την ε, αξιολόγηση την αμοιβαία αξιολόγηση και αν είναι επιτυχής η ιδέα ή όχι. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους γιατί θέλουν ή δεν θέλουν και γιατί πέτυχε ή δεν πέτυχε η αμοιβαία ε, αναγνώριση διότι αν παραβούν τις διατάξεις ε, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπως στη Γερμανία και στη Δανία. Ε, η γερμανική διοίκηση ζήτησε πληροφορίες από την διοίκηση της Δανίας για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην παροχή υπηρεσιών. Αμοιβαία λοιπόν ε, διαδικασία αξιολόγησης, συγγνώμη, είπα αναγνώριση, έκανα λάθος. Αμοιβαία λοιπόν διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία μεταξύ όλων των κρατών μελών και για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι η χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας θα επιβεβαιωθεί όταν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους ενημερώνονται για τις δυσκολίες που υπάρχουν στην παροχή υπηρεσιών. Είναι λοιπόν ε, στο θέμα των Κέντρο αμοιβε... Ε, εξυπηρέτηση, εξυπηρέτησης πολύ σημαντικό να συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε αυτό το θέμα να ολοκληρωθούν τα κέντρα αυτά να αναπτυχθούν να είναι ευκολόχρηστα εύκολα προσβάσιμα και εμείς πιέζουμε τα πέντε κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν έχουν καθόλου αναπτύξει αυτές ε, τις υπηρεσίες ε, ενιαίας, ε, των, των ενιαίων κέντρων, τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Λοιπόν, να συνεχιστεί η πίεση από όλες τις πλευρές να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν τα κέντρα αυτά. Στη διοικητική συνεργασία προσπαθούμε να προχωρήσουμε πρακτικά. Να, ε, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν ε, να συγκεράσουν όλες τις, τις διοικητικές τους υπηρεσίες, να χρησιμοποιούν ε, ε τράπεζες στοιχείων, τράπεζες δεδομένων ευρωπαϊκές, αλλά βεβαίως δεν έχουμε εμείς την εθνική ευθύνη. Τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνα να διοργανώσουν τη διοικητική συνεργασία. Όπως και με τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται αυτά τα κέντρα εάν ας πούμε μια επιχείρηση καθαρισμού γραφείων ή κτηρίων ε, θέλει να εργαστεί σε μια άλλη χώρα, πρέπει να μπορεί να πάρει τις πληροφορίες αυτές. από το ε, κέντρο εξυπηρέτησης. Ε, επανέρχομαι στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και τις πληροφορίες που δεν καλύπτονται. Π.χ. ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι πολύ βασικές πληροφορίες εάν θέλουν επιχειρήσεις να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους πρέπει να πάρουν αριθμό φορολογικού μητρώου. Εάν δεν μπορείς να πάρεις τις πληροφορίες αυτές από πού θα πάρεις τον αφήμι, πού θα αποτανθείς κλπ. Δυσκολεύεται η λειτουργία τους. Πρέπει, έτσι πιστεύουμε στην Κομισιόν, να συνεργαστούμε ρεαλιστικά ώστε οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δεσμευτώ και να πω ότι οι πληροφορίες αυτές οικονομικού περιεχομένου ή δημοσιονομικού περιεχομένου πρέπει να παρέχουν υποχρεωτικά, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το ΦΠΑ και την, ε, όλο το κανονιστικό πλαίσιο του ΦΠΑ στα κράτη-μέλη, εκεί πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να επιτύχουμε μία πρόοδο. Διότι είναι μία πολύ λογική προσέγγιση. Όπως και στο γλωσσικό καθεστώς Υπάρχει, δεν υπάρχει υποχρεωτική παροχή των πληροφοριών σε πολλαπλές γλώσσες, αλλά σιγά σιγά θα γίνει αυτό. Εάν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης θα αυξηθεί και το ενδιαφέρον των επενδύσεων, των διασυνοριακών μετακινήσεων, επιχειρήσεων κλπ. Οπότε σιγά σιγά τα κέντρα αυτά θα παράσχουν τις προφορίες και σε άλλη γλώσσα πλην της του, του κράτους μέλους. Ε, μετά, όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Μάντες για μια ενιαία ηλεκτρονική υπογραφή στην Ευρώπη, θα έλεγα να υποβάλω την ερώτηση αυτή στους συναδέλφους μας ε, στην άλλη διεύθυνση. Η ηλεκτρονική υπογραφή σημαίνει πολλά πράγματα. Όταν αγοράζεται online, ε, δεν θα αναφέρουμε ονόματα τα εκείνων που παρέχουν τις υπηρεσίες χρειάζεται ένα password αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί ασφαλείς υπογραφές τις οποίες εξασφαλίζεται μόνο όταν έχετε ένα πιστοποιητικό που λέει ποιος είστε. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ε, διαβαθμίσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια την ασφάλεια της ηλεκτρονικής υπογραφής. Μπορείτε να έχετε ένα τετραψήφιο password για να αγοράσετε παραδείγματο χάρη βιβλία online. Αλλά για άλλου είδους συναλλαγές χρειάζονται πιο ασφαλείς υπογραφές μπορεί ένα κράτο μέλο να θέλει υψηλότερο, ε, να παρέχει υψηλότερο επίπεδο ε, ασφάλειας. Δεν θα μπορέσουμε να καταργήσουμε όλα τα, τα επίπεδα ασφαλείας ε, επειδή χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Υπάρχει, υπάρχει το θέμα της ηλεκτρονικής περιγραφής περιλαμβάνεται στην ψηφιακή ατζέντα αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όταν χρησιμοποιούνται θα αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη-μέλη και συνεργαζόμαστε σε αυτό, για αυτό το θέμα με τα κράτη-μέλη όπως συνεργαζόμαστε για τα νέα κέντρα εξυπηρέτησης. Κέντρα εξυπηρέτησης. Πάντως, το σχέδιο ε, για την ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο. Κάτι ρώτησε, υπήρξε μια ερώτηση χωρίς μικρόφωνο είναι, ε, ε, η, οδηγία, η οδηγία είναι ευρύ αλλά δεν καλύπτει τα πάντα. Νομίζω άλλωστε ότι υπάρχει ένας ευρωπαϊκός ε, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλά οι συνάδελφοι της Ταξούντ ε, ασφαλώς, ασφαλώς θα είναι διατεθειμένοι να ζητήσουν αυτό το θέμα γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το αφημί. Αλλά ε, είμαι πιο ενημερωμένη για τα θέματα της ε, ηλεκτρονικής υπογραφής. Πάντως πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό το θέμα σε διασυνοριακές, στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Πρέπει λοιπόν να γίνει η κατάλληλη προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και κατάρτιση. Αλλιώς θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση και όπως σας είπα και κατάρτιση. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτε άλλο. Η κυρία ρωτούσε αν ε, καταργήθηκαν αρκετές ε, άδειες, διαδικασίες αδειοδότησης. Υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης της αναλογικότητας των διαδικασιών αδειοδότησης. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα, πάρα πολλοί τομείς που χρειάζονται αδειοδότηση αν πάρουμε, αν πάρουμε παραδείγματος χάρη το παράδειγμα που ανέφερα προηγουμένως με μια εταιρεία ε, καθαριότητας πρέπει να έχει άδεια, ε, να πάρει άδεια προτού αρχίσει να αναπτύσσει δραστηριότητα για να, ότι, να, για να είναι βέβαιο ότι δεν θα χρησιμοποιεί παραδείγματος χάρη τοξικά προϊόντα. Ε, αλλά ορισμένες φορές υπάρχουν απαιτήσει οι οποίες οδηγούν σε διακριτική μεταχείριση και ασκούμε πίεση στα κράτη-μέλη ε, τα ενδιαφερόμενα για να ε, προβούν στις αναγκαίες τροποποίησης. Αν κάτι ξέχασα θα μου το θυμίστε παρακαλώ. Και ακόμα μια φορά συγχαίρω την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ κυρία Μάρτιν Πράτ να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι στο έγγραφο περί πράξης, για την νέα αγορά υπάρχει ένα σημείο που αφορά τη νέα στρατηγική για το ΦΠΑ το 2012 και που προβλέπεται μια αναθεώρηση του συστήματος. Κυρία Ρόιτοβαξ, ζήσατε το λόγο. Εάν έχετε κάτι, το να το πείτε όμως πολύ σύντομα, λακωνικά παρακαλώ. Γιατί πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στην Επιτροπή ε, όταν έδειξε το ζήτημα του ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης. Κατά άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντική πτυχή για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ε, στηρίζω τον ε, σύσταση ενός ε, νέου λόγου, λογοτύπου και θεωρώ ότι τα κέντρα ενός εξυπηρέτησης θα πρέπει να αποτελούν ένα κοινό όραμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τσεχία. Αυτό το ζήτημα παρουσιάστηκε ως μια ευθιέστατη άποψη από τους ε, υπουργούς μας. Ε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και πραγματικά το να μιλήσουν οι υπουργοί για το ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δημιουργία αυτών των ενίων κέντρων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι συνήθω σε προεκλογικέ περιόδους ε, προσπαθούν να δείξουν ότι κάθε καλό προέρχεται από μια εθνική κρατική πρωτοβουλία. Τα εννέα αυτά κέντρα θα πρέπει να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με έναν κατάλογο υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται. Ίσως ε, αυτό να μην έχει πρόθεση ικανοποιητικά μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για την πολύ θετική συζήτηση σήμερα για αυτήν την οδηγία. Βλέπω μία πολύ διαφορετική προσέγγιση από ό,τι στο παρελθόν. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Κοφά ότι δεν θα πρέπει να παίξουμε με να συγκεκριμενοποιήσουμε ορισμένα στοιχεία. Δεν έχουμε δεδομένα τα οποία να μας επιτρέψουν να βγάλουμε συγκεκριμένα ε, συμπεράσματα σήμερα. Δεν έχουμε λοιπόν ακόμα αυτά τα στοιχεία των επιπτώσεων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα στις παρατηρήσεις, ιδιαίτερα ε, ε, σε αυτά που είπε η κυρία Χένσλικ για τα προβλήματα που δημιουργούνται με το σημείο 18 Αυτό το οποίο έγινε στην ε, Γερμανία είναι θα έλεγα γελίο σε ορισμένε περιπτώσεις όπου έπρεπε συγκεκριμένες κοινότητες να κοιτάξουν λεπτομερώς έναν κατάλογο που έπρεπε να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία για το screening, το οποίο, ο οποίος τελικά ήταν αγελίος στις λεπτομέρειες. Ένα άλλο θέμα είναι το άρθρο 2α του αποκλεισμού των εξαιρέσεων από την οδηγία υπηρεσιών δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένος ορισμός αυτών των υπηρεσιών και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που ρωτάν ποια ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ επαγγελματικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών. Ποιες είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχουν οι εργαζόμενοι και ποιες είναι άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή άλλων οργανισμών. Δεν υπάρχει ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τρίτον το άρθρο 2 παράγραφος 2 γιώτα, εδάφιο γιώτα, όπου υπάρχει μόνο το γαλλικό κείμενο. Και, και παραθέτω η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις κοινωνικές υπηρεσίες που αφορούν την κοινωνική στέγαση, τη βοήθεια στα παιδιά και τη βοήθεια στις οικογένειες και τα άτομα που βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά σε κατάσταση ανάγκης που ασφαλίζονται από το κράτος, από παρόχους που έχουν εξοδοτηθεί από το κράτος, από φιλανθρωπικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται ως αυτές από το κράτος. Εδώ λοιπόν αναφέρονται αυτές οι υπηρεσίες και στη Γαλλία και στη Γερμανία έχουν οδηγήσει, έχει οδηγήσει αυτή, αυτό το εδάφιο σε σύγχυση. Διότι ε, προκύπτει το ερώτημα, ε, τι σημαίνει αυτό, παραδείγματο χάρη τα νήπια. Υπάρχουν ε, διάφορες υπηρεσίε μέρημνας, ιδιωτική σταθμή, η εκκλησία έχει παιδικούς σταθμούς, το δημόσιο, Πώς θα χειριστούμε λοιπόν όλες αυτές τις διαφορετικές υπηρεσίες για τα παιδιά, για τα νήπια. Έχει λοιπόν ήδη υπάρξει αυτή η συζήτηση, έχει, έχει ξεκινήσει και δεν νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν και δημιουργούν σύγχυση πρέπει να τα αγνοήσουμε. Υπάρχουν κράτη-μέλη που ακόμα ασχολούνται με αυτό ακόμα δεν έχουν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Οπότε προκύπτει το ζήτημα του τι θα κάνουμε για να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα συγκεχημένα θέματα. Ο κύριος Λόγκεγκάρντ ε, και αυτός με ρώτησε ποια είναι η θέση μου την ενιαία ηλεκτρονική υπογραφή. Εάν κάνετε, υποβάλλετε μια τέτοια πρόταση, εγώ θα την κρίνω θετικά. Πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι πολύ χρήσιμη, ιδίως το θέμα της πρόσβασης στην αγορά. Ε, δεν θα αποφύγουμε αυτό το ερώτημα τι θα κάνουμε με την, ε, το ζήτημα της ενιαίας υπογραφής και δεύτερον τι θα κάνουμε με τον ΦΠΑ. Τουλάχιστον να ξεκινήσει η συζήτηση σε αυτά τα δύο ζητήματα ε, γιατί θα βοηθήσουμε ιδιαίτερα την εσωτερική αγορά. Όσον αφορά το screening στο, μέσα στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Υπάρχει το screening και η διαδικασία του screening και τα δύο είναι θετικά. Ε, μίλησα με έναν δήμαρχο στη Γερμανία και μου είπε ότι προσπάθησα μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας υπηρεσιών να μελετήσω όλες τις διοικητικές λειτουργίες στην υπηρεσία μου Τις εξέτασε λοιπόν όλες ε, τις ε, διοικητικές δουλειές που γινόντουσαν στο Δήμαρχείο του και κατάφερε να τις απλουστεύσει. Όσον αφορά τώρα την αμοιβαία διαδικασία αξιολόγησης, εμένω σε αυτά τα οποία έχω γράψει. Δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα μία μελέτη επίπτωσης της αμοιβαίας αξιολόγησης, γιατί δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Και για το χρονοδιάγραμμα, τέλος, σας θυμίζω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 7 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και η συζήτηση για τις τροπολογίες. Και η ψηφοφορία θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου για να υποβληθεί η έκθεση το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκέπατ. Το επόμενο θέμα δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντεμιά Αμπάντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια συζήτηση η οποία συνεχίζει στην συζήτηση για, τις, ε, για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα μείνουμε λοιπόν σύντομος. Είχαμε μια ανταλλαγή για αυτό το θέμα σε 6 Οκτωβρίου όταν συζητήσαμε για την κοινωνική διάσταση της συνδίκης Λισαβόνας και έλαβα μέρος στις εργασίες ε, της ε, παραταξιακής, ε, διαπαραταξιακής ομάδας για τις υπηρεσίες και στο φόρουμ για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που οργανώθηκαν από την Βελγική Προεδρία που συνεισέφεραν πολλά σε αυτό το τομέα. Ένα μήνυμα σαφές προκύπτει από όλα αυτά, ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε με ρεαλιστικό τρόπο για να ξεπεράσουμε κάποιες ιδεολογικές διαφορές και να εξασφαλίσουμε την προσπελασιμότητα και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Και με αυτό το πνεύμα, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεών μα, είχα υπογραμμίσει την ιδέα ότι οι κοινωνικέ υπηρεσίε γενικού συμφέροντο ε, έχουν μια πολιτική διάσταση, κυρίω σε μια περίοδο οικονομική κρίση. Ενεργούν ω ε, κοινωνικά αμορτισέρ, θα έλεγα, σε περίοδο κρίση. Κατ' επανάληψη, μα έχουν μεταφέρει πολίτε ανησυχίε και υπάρχουν και προβλήματα προβλήματα επικοινωνίας, οι ουσιαστικά προβλήματα που προκύπτουν. Εξού λοιπόν η ιδέα να σκεφτούμε κατά πώ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των κοινωνικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να αξιολογούν καλύτερα αυτέ οι υπηρεσίε, αλλά και να συλλέγουν μια σειρά από πληροφορίε που θα προέρχονται από διάφορε πηγέ στα κρατημένη και θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τι βέλτιστε πρακτικέ είτε είναι ευρωπαϊκέ, εθνικέ ή περιφερειακέ. Έτσι λοιπόν θα δώσουμε μια προβολή πολύ μεγαλύτερη σε αυτές τι κοινωνικέ υπηρεσίε. Το ίδιο επίση ε, ε, στο σελίδα τη Κομισιόν για τις ε, συχνέ ερωτήσεις θα έπρεπε να ε, λειτουργεί στι 23 επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση τη προ του ε, Υπάρχει και η οικονομική προσέγγιση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι γνωρίζετε ότι οι οικονομικέ υπηρεσίε αποτελούν το 9,6% των ε, απασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εργαζόμενοι στι κοινωνικέ υπηρεσίε. Ε, μάλλον και τα ποσά τα οποία θα παρούν στις κοινωνικέ υπηρεσίες καλύπτουν το 9,5 του ΑΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προσέγγιση κατάλληλη ε, και μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Χρειάζεται να σκεφτούμε επίσης και το ζήτημα της ε, διάρθρωσης των ε, αγορών και των κοινωνικών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τους νέους τρόπους διαχείρισης στο πλαίσιο της συνεργασίας δημόσιου-δημόσιου τομέα ή και την περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών κριτηρίων κατά την επιλογή των διαφόρων ε, ε, προμηθειών. Πέραν από την πολιτική και οικονομική διάσταση, οι κοινωνικές υπηρεσίες θα μπορέσουν να ε, επιβιώσουν να συνεχίσουμε να άρουμε μια σειρά από νομικές αβεβαιότητες. Και σας παροτρύνω να εκτάσει το ζήτημα του οδηγού των κοινωνικών υπηρεσιών για τις ε, κρατικές ενισχύσεις και τις ε, προμήθειες δημοσίου. Ο κατάλογος αυτός απαντά σε μια σειρά από ευαιότητες ε, με ενδιαφέρουσες απαντήσεις και θα ήθελα να γνωρίζω λίγο περισσότερο το νομική ισχύ αυτού του καταλόγου. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε να μας διαφωτίσει επί του σημείου αυτού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του νομικού πλαισίου, στο οποίο μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις, ε, γενικές, ε, τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, η έκθεση Μόντι δεν, ε, βλέπει, δεν προσφέρει καμία προσθέμενη αξία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες αυτές με βάση το άρθρο 14 της Συνθήκης Ένωσης, αν και προτείνει να χρησιμοποιούνται σε μια βάση κλαδική. σε όλους τους ε, τομείς ε, που ενέχονται. Τώρα, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια πραγματιστική προσέγγιση, κλαδική προσέγγιση, που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην όλη συζήτηση και να μελετήσουμε μια περίπτωση λογία για να δούμε πώς ε, οι επιπτώσεις αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν και εξηγούμε. Θα ήταν καλό να καλέσουμε την Κομισιόν σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο να κάνει μια σε βάθος έρευνα για τη λειτουργία ενός περισσότερου κλάδου από την τομέα των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Θα μπορούσαμε να εξτάσουμε το ζήτημα των υπηρεσιών παρέχοντα στους ηλικιωμένους που σε ένα πλαίσιο γύρανσης του πληθυσμού θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε μια ακτινογραφία αυτού του κλάδου και να αξιολογήσουμε τι επιπτώσει που έχει στην ε, και θα πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτό τον κοινό στόχο που αφορά την προσβασιμότητα, προσπαλασιμότητα των ε, δημοσίων υπηρεσιών ε, και να αναφερθώ επίσης στην διαφοροποίηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε αυτόν τον κλάδο, διότι η επικουρικότητα παραμένει ένας τομέας που να καθοδηγεί τη σκέψη μα. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη. πρέπει να τηρήσουμε αυτόν τον πλουραλισμό και αυτήν την διαφορετικότητα που υπάρχει και την αποσαφήνιση των ε, διαφορών που υπάρχουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Προς αυτή η κατεύθυνση λοιπόν σας καλώ να προχωρήσετε στο πλαίσιο της όλη της Well, we are pretty, pretty in schedule, late. Έχουμε η ώρα είναι περασμένη. Θέλει κάποιος από του σκιώδει συζητητέ οπωσδήποτε να μιλήσει. Αν ναι, να είναι σύντομο, παρακαλώ. Αν όχι, θα δώσω ένα λεπτό στην Επιτροπή για να μας πει δύο πράγματα. Σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ήδη τη θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα στη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης. Γι' αυτό απλώς θα επαναλάβω ε, θα ε, ε, επανέλθω σε αυτά που μας είπε με πολύ μεγάλη ικανότητα ο κύριος Σαμπάντο, ο οποίος μας έδωσε μια πολύ περιστατωμένη ανάλυση για αυτό το θέμα. Είχαμε άλλωστε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις του στο τελευταίο φόρουμ που οργάνωσε η Βελγική Προεδρία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ε, Επιτροπή η συμμετοχή των διαφόρων επιτρόπων στο φόρουμ και οι εισαγωγικέ παρατηρήσεις του δικού μου επιτρόπου ήταν πάρα πολύ σαφείς. Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών να εφαρμόζουν πιο αποτελεσματικά τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες. Πράγματι, ε, στη διάρκεια του φόρου μοιράσαμε έναν οδηγό ο οποίος ε, απαντά σε πολλά ερωτήματα για την εφαρμογή των κανόνων σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στην εσωτερική αγορά κλπ που αποτελεί μια επικαιροποίηση των ε, ερωτήσεων που είχαν υποβληθεί το 2007. Ο κύριος Αμπάντ ε, ρωτά ποια είναι η νομική αξία αυτών των ε, αποτελεσμάτων. Αυτό είναι είναι ένα έγγραφο που έχει προκύψει από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Μπορούμε λοιπόν να εμπιστευθούμε αυτόν τον οδηγό απόλυτα διότι παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής αυτούς τους κανόνες. Ένας οδηγό, έχει σκοπό να βοηθήσει, βοηθήσει τις εθνικές αρχές να ε, εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες. Είναι πολύ πλήρης είναι πολύ πλήρης αυτός ο οδηγός, διότι έλαβε υπόψη τις ερωτήσεις που λάβαμε για αυτό το θέμα και, τις οποίες, και, και, και τα στοιχεία που πήραμε από τις επαφές που έχουμε με τους εκπροσώπους των κρατών μελών. Και θα ολοκληρώσω ε, λέγοντας κάτι για μια μελέτη που θα μπορούσε να αναλάβει η Επιτροπή, απαντώ στον κύριο Αμπάντ, λέγοντας ότι υπάρχει ήδη μια μελέτη η οποία διεξάγεται ήδη σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς οργανώνονται στην πράξη αυτές οι υπηρεσίες και όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση, με τα χαρά, αν μας το ζητήσετε, θα μοιραστούμε μαζί σας τα αποτελέσματά τη. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς για την υπομονή τους και να πω ότι θα επανέλθουμε ε, σε αυτό το θέμα τον Ιανουάριο, οπότε θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Στις 25 και 26 Ιανουαρίου και ε, η, προθεσμία για την κατάσταση των απολογιών θα είναι στις αρχές Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ και γεια σας.